αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο στη συνεδρίασή του για τον ορισμό υποψηφίου για τη θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διεξήγαγε μία ψηφοφορία κατά την παράθεση για πρώτη φορά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λοιπόν ορίστηκε ως υποψήφιος ο κύριο Jean-Claude Juncker. Κύριε Juncker, σα καλωσορίζω θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα έχετε τώρα τη δυνατότητα να κάνετε την ομιλία σας ε, εν ώψη της διαδικασίας έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Υποψηφιότητας. Σας ε, δίνω το λόγο. Σας ε, χαιρετίζω, χαιρετίζω την παρουσία σας. Λόγω των προηγουμένων ιδιωτήτων σας πολλές ε, είχατε προσέλθει σας συγχαίρω για την υποψηφιότητά σας και σας δίνω το λόγο. Bonjour, Monsieur le Président Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, Στην 25η Μαΐου οι Ευρωπαίοι πολίτες ομίλησαν. Έστειλαν ξεκάθαρα μηνύματα αν και κάπως αντιφατικά. Σήμερα και για τα επόμενα χρόνια εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε, να απαντήσουμε στις προσδοκίες τους, στις αγωνίες τους, στις ελπίδες τους και στα όνειρά τους. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχει θέση και για τα όνειρα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έδρα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας θα παρουσιάσω τους γενικούς προσανατολισμούς της δράσης της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γενικούς προσανατολισμούς επαναλαμβάνω. Περιληπτικά θα τα παρουσιάσω, έτσι και αλλιώς σας έχω στείλει ένα σύντομο κείμενο σε όλες τις επίσημες γλώσσες, γιατί όλες οι γλώσσες την χάνουν της ιδίας αξιοπρέπειας. Να ευχαριστήσω επίσης και τους μεταφραστές οι οποίοι ξενύχτησαν για ένα κείμενο το οποίο τέλειωσα αρκετά αργά χθες το βράδυ. Το λεπτομερές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα ε, νομιμοποιηθεί από τη δική σας ψήφο μετά από την πρόταση του συνόλου των Επιτρόπων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ξεκινάει τώρα διαφέρει από τους προκατόχους του Είστε το πρώτο κοινοβούλιο που ε, πράγματι εκλέγει πράγματι άμεσα κατά κάποιο τρόπο τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια μιας νέας κατάστασης. Είδατε μετά από τις εκλογές ότι έπρεπε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της ε, καθολικής ψηφοφορίας. Έτσι νοηματοδοτήσατε τον δημοκρατικό και τον πολιτικό χαρακτήρα του άρθρου 17, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Χωρίς τη δική σας επιμονή και χωρίς ε, την δική σας προσπάθεια, το άρθρο αυτό θα είχε μείνει γράμμα νεκρό. Προασπιστήκατε λοιπόν τις δημοκρατικές αρχές ε, και είχατε κάθε δίκαιο για να το κάνετε ένα κοινοβούλιο το οποίο επιβάλλει τον σεβασμό της δημοκρατίας ε, κάνει κάτι το σωστό και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να του ασκηθεί κριτική ή να του αποδοθούν άλλου είδους σκέψεις. Θέλω εδώ να ευχαριστήσω και τους ε, υπολείπους ε, υποψηφίους οι οποίοι και αυτοί προσέδωσαν αρκετή ζωηρότητα στην δημοκρατική μορφή διαλόγου. Αν η οικογένεια η πολιτική ενός από αυτούς είχε νικήσει στις εκλογές, είχε κυριαρχεί στις εκλογές, τότε θα ήμουν πρώτος να είναι ο εκπρόσωπος αυτής της ομάδας ο υποψήφιος. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δύο κοινοτικά όργανα, κατεξοχήν θα έλεγα κοινοτικά. Είναι λοιπόν φυσιολογικό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από την άλλη το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να έχουν σχέσεις εργασίας στενότατες. Θα είμαστε κοινοτικοί εταίροι, όχι εναντίον του Συμβουλίου ή εναντίον του Συμβουλίου Υπουργών. Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί εναντίον ή εις βάρος των κρατών και των εθνών δεν είναι μια προσωρινή παρένθεση της ιστορίας αλλά είναι κάτι που διαρκεί στην ιστορία. Εμείς σαν Κοινοβούλιο και Επιτροπή θα δράσουμε προς το κοινό καλό, προς το κοινό συμφέρον και θα το πράξουμε από κοινού. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό δεν καθιστά βέβαια τον Πρόεδρο της Επιτροπής γραμματέα του Συμβουλίου. Η Επιτροπή δεν είναι μια τεχνική επιτροπή από λαμπρούς ανώτατους υπαλλήλους που εξυπηρετεί τα άλλα όργανα. Η Επιτροπή θα είναι ένα πολιτικό όργανο, εγώ θέλω να είναι πιο πολιτική από ό,τι στο παρελθόν και θα είναι. Η σύνθεσή της θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την πολλαπλότητα της πλειοψηφίας η οποία έχει αρχίσει να δημιουργείται στο Κοινοβούλιο και θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν οργανώσει την δική του εσωτερική αρχιτεκτονική να εμπνευστεί από την ίδια αυτή αρχή. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται από το δικό σας σώμα, από τη δική σας ολομέλεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι απλά δέχεται διαταγές. Εγώ δεν θα είμαι ο υπασπιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα πρέπει να αμφιβάλλετε για την επιθυμία μου να θέσω ε, τέλος επίσης στη λειτουργία ενός επιτρόπου από τον οποίο θα αποσύρετε την εμπιστοσύνη σας. Και ταυτόχρονα θα πρέπει αυτά τα οποία ζητάτε, οι παρεμβάσεις σας προς την κατεύθυνση αυτή θα συνοδεύονται από ενέργειες από πλευράς μου. Και το δικαίωμα να θέτετε ερωτήσεις θα παραμένει ελεύθερο όπως λειτουργεί άλλωστε και σήμερα. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τους επιτρόπους να είναι πιο συχνά παρόντες στις σημαντικές τριμερείς συναντήσεις, στους τριμερείς διαλόγους και το Συμβούλιο ελπίζω να κάνει το ίδιο. Ταυτόχρονα το μητρό των λόμπι θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και να καταστεί υποχρεωτικό. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος ήρθε να δει ποιον και νομίζω ότι και τα υπόλοιπα όργανα να μας ακολουθήσουν προς την προσπάθεια αυτή. Je ferai Στόχος μου θα είναι οι κανόνες οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον τομέα σαν παράδειγμα της αδειοδότησης των γενετικά τροποποιημένων να επανεξεταστούν. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ δεν θα έχει διαμορφωθεί προς την κατεύθυνση αυτή μια πλειοψηφία κρατών. Με τον ένα τρόπο ή τον άλλο νομίζω ότι θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις καθαρά ιδεολογικές συζητήσεις οι οποίες δεν δημιουργούν κάτι. Ας τις αντικαταστήσουμε από ειλικρινείς συζητήσεις που οδηγούν σε ισχυρές φιλοδοξίες που θα μας πάνε μακριά. Ας επιλέξουμε όμως τον πραγματισμό σαν μέθοδο. Ας συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες αποφάσεις για να προσφέρουμε στα κράτη-μέλη. Ας μην σταθούμε σε διοργανικές συζητήσεις που μας απομακρύνουν από τον Ευρωπαίο πολίτη. Και θα πρέπει να πω στις κυβερνήσεις ότι θα πρέπει να αντιστέκονται ακόμα πιο πολύ στην πρόθεσή τους να ασκούν κριτική στα ευρωπαϊκά όργανα και σε αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στις Βεξέλλες. Λέτε ναι στις Βρυξέλλες αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πείτε και όχι. και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση μετά από μια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Υπουργών να λέει μια χώρα ότι νίκησε μόνη της εις βάρος των άλλων. Όχι. Στην Ευρώπη ή όλοι νικάμε ή όλοι χάνουμε. Η Ευρώπη έχει καταστεί δυσανάγνωση γιατί πάρα πολύ συχνά μετατρέπουμε την περιγραφή μας σε μια γελιογραφία. Ας μην ομφαλοσκοπούμε εθνικά, ας παίξουμε συλλογικά το παιχνίδι, ας εφαρμόζουμε την κοινοτική μέθοδο. Είναι απαιτητική η μέθοδος αυτή, αλλά έχει αποδειχθεί αποτελεσματική και είναι περισσότερο αξιόπιστη από τις διακυβερνητικές αρνητικές πρακτικές. Πρέπει να αποκατασταθεί η κοινοτική μέθοδος. Αγαπητέ Πρόεδρε, να μιλήσω τώρα στη γλώσσα του παγκοσμίου πρωταθλήτη. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, ναι κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη έχει χάσει αξιοπιστία. Η απόσταση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών έχει αυξηθεί. Μόνο οι κουφή ε, κουφοί και οι τυφλοί δεν το βλέπουν και δεν το ακούν αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά δύσκολα εξηγεί γιατί λειτουργεί. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εξηγούμε γιατί λειτουργούμε στους πολίτες μας. Η Ευρώπη Χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, ένα θεματολόγιο ευραίων μεταρρυθμίσεων. Το status quo δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει. Πρέπει να έχουμε μεταρρυθμίσεις. Πολύ συχνά οι πολίτες φοβούνται όμως τις μεταρρυθμίσεις, διότι θεωρούν ότι μπορεί να τους απειλήσουν, ότι είναι επικίνδυνες. Αλλά όποιος δεν είναι διατεθειμένος να διατρέξει κινδύνους, διατρέχει τον μέγιστο κίνδυνο. Πρέπει να διατρέξουμε κινδύνους, ούτω ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χάσει διεθνή και παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Έχουμε υποχωρήσει γιατί κάναμε σημειωτών. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη κίνηση προς τα μπρος. Η ανταγωνιστικότητα πολύ συχνά ταυτίζεται με μονομερή κατάργηση του κοινωνικού κράτους. Αλλά η ανταγωνιστικότητα δεν επιτυγχάνεται με διάλυση του κοινωνικού κράτους. Η ανταγωνιστικότητα βασίζεται σε ένα τρίπτυχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ενεργό ε, σημείο αναφοράς και για τους πολίτες και για τους εργαζόμενους και για τους επενδυτές. Πρέπει να θυμίσουμε δηλαδή ότι η οικονομία πρέπει να υπηρετεί τους ε, πολίτες και όχι το αντίστροφο. Η οικονομία πρέπει να είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Αυτό μας υποχρεώνει να θεωρούμε ότι οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς δεν μπορούν να προηγούνται των κανόνων για τις ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές. Μόνο μέσω κοινωνικού κράτους θα διατηρήσουμε την εσωτερική αγορά. Είμαι ενθουσιώδης υπέρμαχος της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Ευημερία για όλους, όχι μόνο για λίγους, ευημερία για όλους. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα της οικονομικής και κοινωνικής μας πολιτικής. Πολύ συχνά λέγεται, λόγω της κρίσης, ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς απέτυχε. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν απέτυχε η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Απέτυχαν εκείνοι οι οποίοι στράφηκαν κατά των βασικών αρετών της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για λόγους κερδοσκοπίας. Δεν απέτυχε η κοινωνική οικονομία της αγοράς. Η κοινωνική οικονομία της αγοράς μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν υπάρχει κοινωνικός διάλογος. Ο κοινωνικός διάλογος στα τελευταία χρόνια της κρίσης δεν λειτουργήσε και σε εθνικό αλλά πάνω απ' όλα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να τον αναζωογονήσουμε. Θέλω να είμαι ένας πρόεδρος του κοινωνικού διαλόγου. Πρέπει Επίσης, να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως τόπου παραγωγής. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ανάπτυξη, όχι μέσω αύξηση των ε, χρεών που δημιουργεί καταστροφή. Χρειαζόμαστε βιώσιμη ανάπτυξη για δεκαετίες. Χρειαζόμαστε μια φιλόδοξη πολιτική για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα μέσω επενδύσεων. Γιατί τα χρειαζόμαστε αυτά. Γιατί πολλοί πολίτες στην Ευρώπη θέλουν να επανέλθει η Ευρώπη στο κέντρο της ζωής τους. Τα πακέτα ανάπτυξης, τα πακέτα ανταγωνιστικότητας και τα προγράμματα επενδύσεων έχουν μόνο ένα στόχο. Να βοηθήσουν τους πολίτες να επανέλθουν στο κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτή τη συγκυρία, εντός των ορίων της Ένωσης, υπάρχει ένα 29ο κράτος. Είναι το κράτος των ανέργων. Είναι ένα κράτος στο οποίο κατοικούν οι νέοι άνεργοι, οι αποκλεισμένοι, αυτοί που έχουν μείνει στο περιθώριο της ζωής. Θα ήθελα αυτό το 29ο κράτος μέλος να επανέλθει στα κανονικά κράτη-μέλη. Γι' αυτό έχω ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων να προτείνω. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 θα ήθελα να έχει υποβληθεί αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις. Θα ήθελα τα επόμενα τρία χρόνια να δαπανηθούν 300 δις ευρώ για δημόσιες αλλά κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις. Θα το επιτύχουμε και θα ήμουν ευγνώμων για τη στήριξη του Κοινοβουλίου προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούμε να το επιτύχουμε εάν έχουμε στόχο προσιλωμένη χρήση των υπαρχόντων διαρθρωτικών ταμείων και στόχο προσιλωμένη χρήση και των νέων μέσων που θα δημιουργήσουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για τις υποδομές, χρειαζόμαστε συντονισμένες επενδύσεις, επενδύσεις στον τομέα τον ευρυζωνικό για τα θέματα των ε, ενεργειακών δικτύων, για θέματα επενδύσεων μεταφορών, για κέντρα παραγωγής και βιομηχανίας. Χρειαζόμαστε μια επαναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στο βιομηχανικό τομέα. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για την έρευνα, την ανάπτυξη, βιώσιμες, ε, ανανεώσιμες ενέργειες. Οι ανανεώσιμες ενέργειες δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν καλές προθέσεις στην οικολογία. Η ανάπτυξη των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας είναι προϋπόθεση ούτως ώστε η Ευρώπη να έχει μόνιμη βιώσιμη ανάπτυξη που θα κατοχυρώσει την ε, οικονομική της θέση στον κόσμο. Μια Ευρώπη που θα επενδύει είναι μια Ευρώπη που θα ευημερεί. Μια Ευρώπη με περισσότερη απασχόληση. Οι επενδύσεις είναι ο καλύτερος σύμμαχος των ανέργων. Παράλληλα, πρέπει να λειτουργήσει και να επεκταθεί περισσότερο το σύστημα εγγυήσεων για την ανεργία των νέων. Θα ήθελα σταδιακά να περάσει από τα 25 στα 30 χρόνια. Οι επενδύσεις μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εάν μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Κυρίως όσον αφορά τις μικρομέσαες. Οι μικρομεσαίες δεν είναι οι μεγάλοι καπιταλιστές. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δουλεύουν μέρα νύχτα, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να έχουμε αποφασιστική μείωση της γραφειοκρατίας. Των γραφειοκρατικών υπερβολών. Πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά την αρχή της επικουρικότητας. Από τη συνθήκη του Μάστρικ και εντεύθεν συζητάμε για τη σωστή χρήση και εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Αλλά δεν την εφαρμόζουμε παρά μόνο πλημελώς. Και οι προσπάθειες για την κατάργηση της γραφειοκρατίας πρέπει να συνδυαστούν με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Δεν χρειάζεται να αναμειγνύονται σε όλες τις λεπτομέρειες ε, της ε, οικονομικής δραστηριότητας. Πρέπει να ασχολούνται με τα κύρια προβλήματα της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν κάθε πρόβλημα ωστόσο που υπάρχει στην Ευρώπη να είναι πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα κυριότερα θέματα. Όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, πρέπει φυσικά να ε, συμβαδίζουν με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν θα τροποποιηθεί όσον αφορά τις βασικές του κατευθύνσεις. Αυτό το καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα βασιστώ τα επόμενα χρόνια σε αυτές ακριβώς τις καθευντήριες γραμμές. Και την σταθερότητα μας την υποσχέθηκε η εισαγωγή του κοινού νομίσματος. Αλλά η σταθερότητα πρέπει να ισχύει πάντα. Αυτήν έχουμε υποσχεθεί. Και η Ευρώπη πρέπει να τηρεί τις υποσχέσεις της. Και δεν θα τις ε, διαψεύσω εγώ. Αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σωστά διαπίστωσε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε το περιθώριο ευελιξίας που περιέχει το Σύμφωνο Σταθερότητας μετά τις πρόσφατες τροποποίησεις του, ούτως ώστε η διάσταση ανάπτυξη του συμφώνου αυτού να μπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως. Το κάναμε και στο παρελθόν αυτό. Θα το κάνουμε και στο μέλλον περισσότερο. Οπότε έρχομαι στη διαπίστωση κύριε Πρόεδρε ότι αυτά που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια αυτά που επιτύχαμε δεν θα πρέπει να υποτιμούνται. Ήμουν πρόεδρος ε, του Eurogroup και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν ε, ψυχαγωγία. Νομίζω ότι υπάρχουν πολύ ε, ε, πιο ευχάριστα αξιώματα από αυτό. Αλλά κατά την ε, κρίση του, για την ευρωκρίση που δεν ήταν κρίση του ευρώ αλλά κρίση χρέους, καταφέραμε να επιδιορθώσουμε εν πτήση ένα φλεγόμενο αεροσκάφος. Δεν ήταν απλό. Χρειαζόταν μεγάλη τέχνη που μπορεί, βεβαίως αυτό που κάναμε μπορεί να μην ήταν πάντα, πάντα, πολύ ε, μεγάλη δεξιοτεχνία, αλλά παρόλα αυτά το καταφέραμε. Ξέρετε ότι για χρόνια κερδοσκόποι διαφόρων ε, προελεύσεων και πολύ ε, με χερεκακία προέβλεπαν ότι θα κατέρευε η Ευρωζώνη, αλλά δεν, δεν κατέρευσε. Σε πολλές χρηματαγορές έγιναν στοιχήματα ότι η Ελλάδα θα εξέρχεται από την Ευρωζώνη. Έκανα ό,τι μπορούσα και είμαι περήφανος που η Ελλάδα αυτή, αυτό το μεγάλο έθνος, αυτός ο θαυμάσιος λαός εξακολουθεί να είναι μέλος της Ένωσής μας. Aber, Herr Präsident, wir haben noch Fehler gemacht. Αλλά κάναμε και λάθη κύριε Πρόεδρε. Ένα φλεγόμενο αεροπλάνο εν πτήση δεν διορθώνεται εύκολα από καιρό καιρό, από καιρούς καιρό ε, καίγεται και λιγάκι κανείς. Πιστεύω ότι στο μέλλον όταν θα έχουμε προγράμματα προσαρμογής και ελπίζω να μην υπάρξει στο μέλλον αυτό, θα ήθελα λοιπόν πριν χρειαστούν προγράμματα προσαρμογής θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες κοινωνικές μελέτες. Θα ήθελα να ξέρουμε πώς ακριβώς ε, λειτουργεί και τι επιπτώσεις έχουν τα προγράμματα προσαρμογής στη ζωή των ανθρώπων χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων ανάλυση των πολιτικών επιπτώσεων δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται προγράμματα προσαρμογής. Και επίσης θα ήθελα κάθε φορά που εκπονούμε πρόγραμμα προσαρμογής να έχουμε και μία εναλλακτική λύση, ένα σχέδιο Β που να μπορούμε να το εφαρμόσουμε όταν οι μακροοικονομικές συνθήκες δεν ισχύουν για το σχέδιο Α, όταν υπάρχει λιγότερη ανάπτυξη από αυτήν που είναι η βάση του προγράμματος προσαρμογής. Τότε θα πρέπει να προσαρμόζονται ακριβώς τα προγράμματα προσαρμογής. Γι' αυτό θα πρέπει, θα πρέπει να έχουμε έτοιμο και ένα εναλλακτικό σενάριο. Α, δεν σας πείθει. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης να ξανασκεφτούμε το μέσον Τρόικα. Το Κοινοβούλιο υπέβαλε τη σχετική έκθεση όπου λέει ότι λείπει δημοκρατική ουσία από τον τρόπο λειτουργίας της Τρόικα. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική διάσταση. Θα πρέπει να επαναδιαμορφώσουμε την Τρόικα, ούτως ώστε να είναι πιο δημοκρατική, πιο πολιτική, πιο κοινοβουλευτική. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να δαπανάμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Πρέπει να αντικαταστήσουμε όμως ε, το χρέος με ιδέες. Οι ιδέες υπάρχουν. Πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει η ψηφιακή τεχνολογία η οποία δεν γνωρίζει σύνορα. Πρέπει να ξαναδούμε τις ρυθμίσεις για τις τηλεπικοινωνίες, για το copyright, για την προστασία δεδομένων πρέπει να δούμε ξανά τι ισχύει στις χώρες μέλη για όλα αυτά. Δεν πρέπει να βάζουμε σύνορα σε αυτά. Πρέπει, πρέπει να εξαφανιστούν τα τέλη περιαγωγής συνολικά στην Ευρώπη. Πρέπει για να είμαστε επιτυχείς να εφαρμόσουμε μια πραγματική ψηφιακή αγορά με 250 δισεκατομμύρια επιπλέον ανάπτυξη για την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει επίσης, όπως έχει υποθεί τόσο συχνά, κυρίως κατά τη διάρκεια της Ουκρανικής κρίσης, χρειαζόμαστε μια πραγματική ενεργειακή ένωση και αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών με την κατάλληλη πολιτική μας. Πρέπει να επαναδιοργανώσουμε την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτήσουμε μια νέα ενεργειακή ένωση στην Ευρώπη. Να βάλουμε μαζί τις δυνατότητες που έχουμε, τους πόρους που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε ε, την κατάσταση σε σχέση με τρίτες χώρες. Πρέπει να αποφεληθούμε από τους ενεργειακούς πόρους που διαθέτουμε και να βελτιώσουμε την ενεργειακή αυτονομία των χωρών μελών μας. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση θα γίνει αριθμός ένα στον κόσμο και θα ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή αυτονομία και τους στόχους του 2020. Πρέπει να έχουμε ένα δεσμευτικό ποσοστό 30%. Για μένα αυτό είναι το ελάχιστο μάλιστα αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Βλέπετε δεν είναι δυνατόν να μην είμαστε στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο εφόσον έχουμε ενεργειακή αυτονομία. Η εσωτερική αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί, να είναι πλήρης. Αν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε άλλα 200 δισεκατομμύρια στην ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να συμπληρώσουμε λοιπόν τους νέους κανόνες για τις τράπεζες με την ε, νέα κεφαλιακή αγορά. Πρέπει να βελτιώσουμε τις οικονομίες μας και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε νέες ολοκληρωμένες ε, κεφαλαϊκές αγορές. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε εφόσον υπάρξουν περισσότερα κεφάλαια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων τώρα πάντα ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της εσωτερικής αγοράς. Θα στηρίξω λοιπόν αυτή την αρχή. Η ελεύθερη διακίνηση δεν είναι μόνο μια ευκαιρία. Δεν θα αλλάξουν οι κανόνες. Είναι οι, οι χώρες μέλη οι οποίες θα αποφασίσουν παρετέρω για τις ρυθμίσεις τους. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι ότι θα προσπαθήσουν να δούμε και πάλι την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και το πώς αυτή εφαρμόζεται. Πρέπει να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ και θα το κάνουμε. Το θέμα της φοροδιαφυγής επίσης είναι ένα θέμα που επίσης θα κοιτάξω και θα ήθελα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει υιοθέτηση ενός κειμένου που να έχει να κάνει και με τις ε, οικονομικές συναλλαγές. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος και θα το κάνουμε. Όσον αφορά τώρα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω εδώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι η κρίση δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει η κρίση. Δεν τελειώνει η κρίση όσο υπάρχουν τόσοι άντρες και γυναίκες που βρίσκονται στην ανεργία. Όσο δεν έχουμε την πλήρη απασχόληση δεν θα έχει τελειώσει η κρίση. Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα τις οικονομικές μας πολιτικές. Πρέπει να έχουμε μια οικονομική διακυβέρνηση, κάποιου είδους οικονομική κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο και θα το κάνουμε πρέπει να παραμείνουμε απαιτητικοί όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες και θα συνεισφέρουν στην οικονομική μεγέθυνση στην Ευρώπη. Εάν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης κάνουν παραπάνω προσπάθειες, πρέπει και εμείς να βρούμε τα οικονομικά κίνητρα τα οποία θα βοηθήσουν τη διαδικασία αυτή. Και σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να σκεφτούμε την ε, δημιουργία ενός ειδικού προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Πρέπει να δούμε επίσης πώς εκπροσωπούμεθα εμείς που έχουμε ένα από τα πιο ισχυρά νομίσματα στον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να μην υπάρχουν αντιφάσεις, αλλά αντίθετα η Οικονομική και Νομισματική Ένωση να ενισχυθεί και το ευρώ να εκπροσωπείται με μία φωνή, με μία θέση, με μία καρέκλα. Bretton Woods, στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω λοιπόν και δύο λόγια για τη συμφωνία μας ε, ελεύθερων συναλλαγών ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ θα ήθελα να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή. Πιστεύω ότι πρόκειται για τους μεγαλύτερους οικονομικούς χώρους στον κόσμο και για τις μεγαλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο. Οπότε είναι προς το συμφέρον και των Αμερικανών και των Ευρωπαίων να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή. Όμως δεν θα ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή με οποιοδήποτε τίμημα. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε τις δικές μας αρχές στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, ούτε θα εγκαταλείψουμε τις δικές μας αρχές στον κοινωνικό τομέα. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τις δικές μας απαιτήσει όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Δεν θα ήθελα η προστασία των δεδομένων να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς φίλους μας. Και δεν θα ήθελα να έχουμε παράλληλες ε, δικαιοδοσίες. Εμείς είμαστε ένας χώρος δικαίου και εμείς στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζουμε το δίκαιο και να φροντίσουμε οι διαπραγματεύσεις αυτές να γίνονται με όσο γίνεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχω να σας πω το εξής. Αν δεν δημοσιεύουμε τα σχετικά έγγραφα εδώ μιλάω για τη στρατηγική βέβαια της διαπραγμάτευσης, όχι, αλλά για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Αν δεν υπάρχει διαφάνεια σε αυτό, τότε θα αποτύχουμε. Και εδώ στο Κοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια η συμφωνία αυτή θα αποτύχει αν δεν υπάρχει τέτοια διαφάνεια. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Στο κάτω-κάτω δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι κάτι θέλουμε να κρύψουμε. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών. Είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και είμαστε αξιόπιστοι αν είμαστε απαιτητικοί στο θέμα των δικών μας θεμελιωδών αρχών και αξιών. Θα υπάρξει ένας επίτροπος ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο γίνεται πιο γρήγορα να προχωρήσει και στην Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Θα προσπαθήσω επίσης να πείσω το Συμβούλιο να εγκρίνει τη σύμβαση αυτή όσο γίνεται πιο γρήγορα, τουλάχιστον στις κύριες κατευθυντήριες γραμμές. Έρχομαι τώρα στην μετανάστευση νόμιμη, παράνομη. Αυτά είναι θέματα τα οποία σε καθημερινή βάση απασχολούν τους συμπολίτες μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κοινή πολιτική στο άσυλο και θα προτείνω μια τέτοια κοινή πολιτική ασύλου. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό στην Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια της, γιατί τη χρειαζόμαστε. Όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδάς, η Αυστραλία, έτσι και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παρέμβαση στην αίθουσα εκτός μικροφώνου. Ναι, το φανταζόμουν, λέει ο κ. Γιούγκερ, ότι θα υπήρξαν τέτοιες στιγμές ε, έντασης, και ήξερα ότι θα είναι σε αυτό το σημείο της ομιλίας μου. Λοιπόν, να προστατεύουμε τα εξωτερικά μας σύνορα. Να καταπολεμήσουμε τις συμμορίες αυτές που βγάζουν χρήματα από τις ζωές των άλλων. Και ας φροντίσουμε για αυτούς πριν πάρουν τις σχεδίες στα σκάφη να έρθουν στις χώρες μας. Να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεγγύη ανάμεσα στο βορρά και το νότο της Ευρώπης. Η παράνομη μετανάστευση, οι πρόσφυγες δεν είναι προβλήματα της Μάλτας, της Κύπρου, της Ιταλίας, είναι ολόκληρης της Ευρώπης προβλήματα. Äh, Για την εξωτερική πολιτική κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πω πολλά. Η εξωτερική πολιτική, μια κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας είναι κάτι που χρειαζόμαστε επιγόντως. Και θα κάνω αυτό που χρειάζεται ούτως ώστε να μην ε, τροχοπεδείται ο ύπατος εκπρόσωπός μας από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Θα πρέπει να έχει αυτονομία ο ύπατος εκπρόσωπός μας για εξωτερική πολιτική. Εκείνος ή εκείνη που θα αναλάβει αυτό το αξίωμα θα πρέπει να έχουν ένα ευρύ πλαίσιο εργασίας και θα πρέπει να βοηθούνται από τους άλλους επιτρόπους ε, που θα έχουν αρμοδιότητες ε, σχετικές διότι στόχος μας δεν είναι να είναι αντίπαλος του ΝΑΤΟ η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να συνεργαστούν οι δύο αυτοί, να εργάζονται από κοινού. Αλλά στον τομέα της συνεργασίας χρειαζόμαστε περισσότερη ενισχυμένη συνεργασία όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και πάνω απ' όλα τη χρειαζόμαστε στον τομέα των προμηθειών δεν είναι δυνατόν η πολιτική μας για αμυντικές προμήθειες να γίνεται ανταγωνιστικά μεταξύ των κρατών μελών. Κύριε Πρόεδρε, τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα πέντε χρόνια, δεν θα υπάρξει ε, καμία περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης. Από την ε, ε, τωρινή συγκυρία όπως είναι, δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι ε, κάποια υποψήφια χώρα ε, θα μπορέσει να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις ε, μέχρι το 2019. Αλλά οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και έθνη χρειάζονται μια αξιόπιστη, ειλικρινή ευρωπαϊκή, πολιτική, ε, ευρωπαϊκή προοπτική. Αυτό ισχύει κυρίως για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είχαν μια τόσο πρόσφατα τραγική ιστορία και γι' αυτό χρειάζονται μια ευρωπαϊκή προοπτική για να ξεπεράσουν αυτή τη φάση της ιστορίας τους. Θα ήθελα να επανέλθω και στα θέματα της απαραίτητης βιομηχανικής πολιτικής για την Ευρώπη. Απαραίτητης λέγω έτσι ώστε να αυξηθεί και το ε, ευρωπαϊκό ακαθάριστο και να φτάσει το 20% το τμήμα της βιομηχανικής παραγωγής. Θα ήθελα να σας μιλήσω επίσης ε, και την, για, για την Ουκρανία, να χαιρετήσω τον Ουκρανικό λαό, ένα ευρωπαϊκό λαό που έχει τη θέση του στην Ευρώπη. Θα ήθελα να σας εξηγήσω και με περισσότερες λεπτομέρειες γιατί πιστεύω ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρξουν ελάχιστα κοινωνικά εισοδήματα, εγγυημένα ελάχιστα κοινωνικά εισοδήματα Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε κάποια φάση. Αλλά θα ήθελα να πω ότι οι καθολικού τύπου υπηρεσίες και οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρηθούν. Δεν θα πρέπει να αφαιθούν στο έλεος της αγοράς. Πρέπει να υπερασπιστούμε τις δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα επίσης να σας μιλήσω και για την Αφρική για μια τόσο δυστυχή πολύ συχνά Αφρική, για μια τόσο ξεχασμένη Αφρική αλλά τόσο πλούσια Αφρική, Αφρική πλούσια και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Να σταματήσει αυτό το σκάνδαλο, αυτό το δράμα, αυτή η τραγωδία κάποιος πεθαίνει κάθε έξι δευτερόλεπτα από την πείνα και χάνουμε την ημέρα 25.000 παιδιά από την πείνα. Λοιπόν, όσο αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει, η Ευρώπη δεν τελείωσε. Η Ευρώπη είναι υπεύθυνη. Η Ευρώπη συνεχίζει. Ε, θα πρέπει να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να ακούσουμε αυτούς που μίλησαν στις 25 Μαΐου. Αλλά δεν ήρθε η ώρα της Επανάστασης, αλλά ούτε και της αντεπανάστασης. Αν θέλουμε οι Ευρωπαίοι να αγαπήσουν για μια ακόμη φορά την Ευρώπη, να τους πούμε ότι είμαστε υπερήφανοι για την Ευρώπη, να τους πούμε ότι είμαστε περήφανοι για πολλά από αυτά που πετύχαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Λέμε συχνά ότι το θέμα του πολέμου και της ειρήνης δεν τίθεται πλέον, όμως όχι και ιδιαίτερα θα έλεγα ενάρετος διάλογος ανάμεσα στην, στον πόλεμο και στην ειρήνη φαίνεται ότι εξακολουθεί να είναι μια απειλή ε, ιδιαίτερα αν δει κανεί το τι συμβαίνει στα εξωτερικά μας σύνορα. Ας είμαστε περήφανοι επίσης και για τις παλιότερες γενιές οι οποίες έδωσαν τη μάχη τους και ιδιαίτερα μετά από το δεύτερο πόλεμο και μετά από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν για να είμαστε εμείς εδώ σήμερα. Τους το οφείλουμε. Να είμαστε περήφανοι επίσης γιατί στη δεκαετία του 90 πετύχαμε την διεύρυνση μπορέσαμε να συνδυάσουμε την ιστορία και τη γεωγραφία στην Ευρώπη. Ε, τερματίσαμε τη διέρεση, τη μεταπολεμική της Ευρώπης. Ξεπεράσαμε τη λογική αυτή. Χωρίς όπλα, αλλά με πεπιθήσεις, με ιδέες, φέραμε κοντά ιστορικά και γεωγραφικά. Να συγχαρώ λοιπόν για μια ακόμη φορά αυτούς που στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη αποφάσισαν να πάρουν την ιστορία στα χέρια τους. Να μην υφίστανται την ιστορία αλλά να γράψουν μόνοι τους την ιστορία. Ας μην μιλάμε λοιπόν για παλιά μέλη και για νέα μέλη. Υπάρχουν τα κράτη-μέλη, ούτε παλιά ούτε καινούργια. Et soyons και ας είμαστε τέλος υπερήφανοι που δημιουργήσαμε το ενιαίο νόμισμα. Το ενιαίο νόμισμα δεν διαιρεί την Ευρώπη, το ενιαίο νόμισμα προστατεύει, προστατεύει λέω την Ευρώπη. Ήμουν υπουργό οικονομικών στη χώρα μου για 20 χρόνια. Κάθε 6 μήνες έπρεπε να πηγαίνω στις Βρυξέλλες και να είμαι παρόν ε, σε ε, αλλαγές σε επίπεδο συναλλαγματικών αλλαγών. Πραγματικά υπήρχε μια τρομερή αταξία νομισματική, επικίνδυνη αταξία για την ευρωπαϊκή οικονομία. Επανειλημμένα έζησα δύσκολες στιγμές την απώλεια της αξιοπρέπειας μιας χώρας που επειδή δεν μπορούσε να παραμείνει ανταγωνιστική έπρεπε να μειώσει την αξία του νομίσματός της, να υποτιμήσει το νόμισμα της. Με πικρία ήμουν μάρτυρα σε τρομερές σκηνές αυτοί που έπρεπε να υπερτιμήσουν το νόμισμά τους δεν ήθελαν να το κάνουν γιατί φοβόντουσαν τις αγορές και αυτοί που ήθελαν να υποτιμήσουν δεν το έκαναν επίσης γιατί φοβόντουσαν ότι θα υπήρχε μια άτακτη επιστροφή του πληθωρισμού. Αν κατά τη διάρκεια αυτών που συνέβησαν στην Ουκρανία, αν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης την οποία βιώσαμε, και γίναμε το επίκεντρο μιας μεγάλης μάχης. Αν ήμασταν στο παλιό σύστημα τότε η Ευρώπη σήμερα θα ήταν σε πόλεμο. Η Γαλλία εναντίον της Γερμανίας, η Γερμανία εναντίον της Ιταλίας, η Ιταλία εναντίον της Ισπανίας, όλοι εναντίον όλων. Η Ευρώπη λοιπόν, η πειθαρχία της Ευρώπης και οι φιλοδοξίες της Ευρώπης την καθιστούν έναν προστατευτικό οικονομικό πόλο. Και η Ελλάδα κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα δεν ήθελε να εγκαταλείψει την νομισματική ζώνη και δεν θέλαμε κι εμείς να γίνει κάτι τέτοιο. Και τι γίνεται με το Ηνωμένο Βασίλειο, τι γίνεται με τη Μεγάλη Βρετανία, απαντά ο πρόεδρος Γιούνκερ. Εγώ είμαι υπέρ του ενιαίου νομίσματος γιατί προστατεύει την Ευρώπη, την οικονομία της και τους πολίτες της. Κύριε Πρόεδρε, αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα οποία κάναμε τις τελευταίες δεκαετίες, αν δεν είχαμε καταστήσει την Ευρώπη μια ειρηνική Ευρώπη, αν δεν είχαμε συμφιλιώσει την ιστορία και τη γεωγραφία, αν δεν είχαμε δημιουργήσει το ενίο νόμισμα και αν δεν είχαμε οικοδομήσει τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά, σκεφτείτε σε τι κατάσταση θα βρισκόμασταν σήμερα. Σκεφτείτε λίγο. Θα ήμασταν πραγματικά χωρίς όπλα, θα ήμασταν εξασθενημένοι, θα είχαμε προβλήματα, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα. Χάρη στην προσπάθεια των προκατόχων μας η Ευρώπη σήμερα είναι μια ήπειρος η οποία έχει κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη να ζουν στην ειρήνη και στην ευημερία. Κύριε και μια στιγμή, μια στιγμή. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας καταλαβαίνουμε και όταν δεν φωνάζετε τόσο πολύ. Λίγο πιο σιγά. Δεν είναι αναγκαίο μονίμως να διακόπτε τον ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, δεν θέλω μια Ευρώπη η οποία να μένει στάσιμη. Δεν θέλω μια Ευρώπη η οποία να παρατηρεί τους άλλους για το τι κάνουν, για το πώς δρούνε κτλ. Δεν θέλω να είμαι μόνο ένας θεατής. Θέλω μια Ευρώπη η οποία να βρίσκεται στο κέντρο, η οποία να προχωράει, να κερδίζει, να προστατεύει, να υπάρχει. Θέλω μια Ευρώπη που να αποτελεί μοντέλο για τους υπόλοιπους, πρότυπο. Και για να το πετύχουμε αυτό, ας εμπνευστούμε από αρχές και πεπιθήσεις που μας ε, κληρονόμησαν οι μεγάλοι Ευρωπαίοι τότε που εκείνοι βρισκόντουσαν στην πρώτη γραμμή όταν εμείς δεν υπήρχαμε ακόμα. Ο Ντελόρ πρώτα απ' όλα, ο μεγάλος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Ζακ Ντελόρ. Ο Ντελόρ είναι φίλος μου και θα εμπνευστώ από το δικό του το έργο. Εδώ θέλω να θέσω και αφορώ τιμή στον Φρανσό Μιτεράν. Ο Μιτεράν ο οποίος είπε ότι οι εθνικισμοί οδηγούν στον πόλεμο. Είχε δίκιο ο Μιτεράν. Θέλω επίση να αποθέσω φόρο τιμή στον Χέλμουντ Κόλ, ο οποίος για μένα ήταν ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος τον οποίο γνώρισα. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμά τους. Είχαν υπομονή, θάρρος, αποφασιστικότητα. Ας έχουμε και εμείς το ίδιο θάρρος, την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια υπομονή. Αυτά τα τρία επιβάλλονται όταν κανείς έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να κάνουμε πολλά μεγάλα πράγματα μαζί για την Ευρώπη, για τους πολίτες της, για τον κόσμο ολόκληρο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιούγκα. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στους Προέδρους των ομάδων και τους εκπροσώπους των μη γεγραμμένων. Οπότε πρώτος για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο κύριος Δίμπα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Ζωάν Γιούγκα, σήμερα είναι μια καλή μέρα για την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα απέδειξαν τις τελευταίες εβδομάδες ότι έχουμε κάθε δυνατότητα να δράσουμε. Οι πολίτε κατά τι ευρωεκλογέ ψήφισαν για το μέλο Ευρώπη για περισσότερη δημοκρατία για μεταρρυθμίσει ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργεί, παρά τι κοινωνικέ επιπτώσει τη μεγάλη χρηματοπιστωτική χρήση. δημιουργήσαμε μια πλειοψηφία επικοδομητική που θα διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρώπη με αυτές τις εκλογές ε, επέτυχε μια μεγάλη δημοκρατική νίκη. Είναι ιστορική μέρα σήμερα. Για πρώτη φορά οι εκλογείς αποφάσισαν για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συναποφάσισαν. Αυτό δεν το επέτυχε ο καθένας μόνος του αλλά, και δεν είναι τα πάντα, αλλά είναι μια σημαντική αρχή. Η αρχή αυτή του επικεφαλής ψηφοδελτίων μπορεί να θεωρείται καλή ή κακή από διαφόρους, αλλά για ένα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι καλύτερα να πούμε από τους να πούμε στους εκλογείς πριν από τις εκλογές τι θέλουμε και με ποιους θέλουμε να κάνουμε κάτι και όχι να το λέμε μετά τις εκλογές. Επί της αρχής αυτής βασιστήκαμε για να επιτύχουμε κάτι. Και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν θα μπορέσει να το ακυρώσει. Είναι καλή μέρα λοιπόν για την Ευρώπη και ως πρόεδρος πολιτικής ομάδας πρέπει να πω ότι είναι μια καλή μέρα και για την πολιτική μου ομάδα και για το κόμμα μου. Έχουμε εδώ τον υποψήφιο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να τον ψηφίσουμε. Για την Προεδρία της Επιτροπής θέλω να, υπενθυμίσω σε όλες τις ε, χώρες ε, που ε, ε, υπέστησαν προγράμματα προσαρμογή. Θέλω να επιθυμίσω ότι όλε αυτέ οι χώρε έχουν αυτή τη στιγμή κυβερνήσει του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Βεβαίω ε, υποχώρησαν οι κοινωνικέ κατακτήσει, αυξήθηκαν οι φόροι, πολλά δυσάρεστα χρειάστηκε να εξηγήσουμε στου πολίτε. Ζητήσαμε πολλά από του πολίτε. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσει αυτέ απέδειξαν στο Λουξεμβούργο, στην ε, Γερμανία, στη Φιλανδία ότι μπορούν να εκφράσουν την αλληλεγγύη την αλληλεγγύη τους στις ε, προεκλογικές εκστρατείες. Όλα αυτά που κάναμε υπέστησαν κριτική από πολλούς. Αλλά εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ υπερασπιστήκαμε αυτές τις αποφάσεις και εξηγήσαμε στους πολίτες γιατί ήταν αναγκαίες. Δεν ήταν απλό, αλλά παρόλα αυτά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επανεξελέγει ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ κέρδισε τις εκλογές. Είναι ο σωστός υποψήφιος τη σωστή στιγμή. Ο Ζαν Κλοντ-Γιούγκερ είναι υποψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ναι, αλλά σήμερα θα υπερψηφιστεί από το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρουμε ότι η αρχή της δημοκρατίας είναι η συμβιβασμοί. Και οι απόψει των άλλων επικοδομητικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνουν ακουστέ. Ο Ζαν Κλοντ Κλοντ-Γιούγκερ εξελέγει με βάση το πρόγραμμα του ΕΛΚ, αλλά στόχο του είναι να επιτευχθεί συνένεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό θα υποστηριχθεί και από τη δική μας πολιτική ομάδα. Λοιπόν, από τη δική του πολιτική ομάδα υπόθηκαν πολλά για μεταρρυθμίσεις μια νέα αρχή. Είναι σαφή τα καθήκοντά μας. Ε, περιγράψαν σαφώς. Για το ΕΛΚ τα επόμενα τέσσερα σημεία είναι τα εξή. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, η Ευρώπη πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Χρειαζόμαστε επαναβιομηχάνηση της Υπήρου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερον, πρέπει να υποστηρίξουμε την σταθερότητα. Τα χρέη δεν δημιουργούν σταθερότητα, δεν καταστρέφουν. Τρίτον, χρειαζόμαστε περισσότερο σεβασμό για τα εθνικά επίπεδα, ιδιαίτερα για τους ε, συναδέλφους μας στα εθνικά κοινοβούλια. Και τέταρτον, μετά τα έτη της κρίσης, η Ευρώπη πρέπει να στραφεί και πάλι προς τα έξω για την πολιτική προσφύγων ή για τις εταιρικέ σχέσεις με τους φίλους μας στην Ουκρανία. Αυτές οι τέσσερις προτεραιότητες τις οποίες ε, υπογραμμίζω στηρίζει το ΕΛΚ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα ε, εξηγήσω ε, λεπτομεριακά την πολιτική μας. Σήμερα θα αξιοποιήσω το χρόνο ομιλίας για να ε, εκφράσω δύο βασικά θέματα για τον πολιτισμό και το πώς αντιμετωπίζουμε την Ευρώπη. Καταρχάς, να, αναφέρω κάποια σημεία που ανέφερε και ο Ζαν Κλοντ Όταν μιλάμε για αλλαγές, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι για πολλούς συμπολίτε μας ε, οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές ε, θεωρούνται απειλητικές. Φοβούνται οι συμπολίτε μας τις αλλαγές. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να κερδίσουμε τους συμπολίτε μας για αυτές τις μεταρρυθμίσεις, για αυτές τις αλλαγές. Πρέπει να έχουμε κάθε συνείδηση ότι σήμερα είμαστε σε μια συγκυρία όπου υπάρχουν πολλές θεμελιώδεις αλλαγές. Πριν από 100 χρόνια η βιομηχανοποίηση ήταν ε, η βασική αλλαγή που δημιούργησε και τότε βεβαίω ε, κερδισμένους και χαμένους, αλλά άλλαξε την κοινωνία. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου γίνονται θεμελιώδεις αλλαγές, πολύμορφες που ποτέ πριν δεν είχαν συμβεί. Σκεφτείτε τις δημογραφικές αλλαγές. Σήμερα έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό άνω των 65. Το 2050 δεν θα είναι 15% όπως σήμερα, αλλά 25% αυτοί που είναι πάνω από 65. Όλα αυτά θα τροποποιήσουν την Ήπειρό μας. Σκεφτείτε επίσης την παγκοσμιοποίηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ευημερία ανακατανέμεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Ο ρόλος της Ευρώπης γίνεται μικρότερος. 24 χρόνια το 2040 δεν θα υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό κράτο στο G7 με βάση τι οικονομικέ του διαστάσει. Αυτό νομίζω ότι είναι εύκολο το στοιχείο. Σκεφτείτε την κλιματική αλλαγή, την οικολογία, το θέμα τη ψηφιακοποίηση. Πώ ε, ερχόμαστε σε επαφή με του φίλου μα, πώ ε, κάνουμε τι αγορέ μα. Όλα αλλάζουν μέσω τη ψηφιακή οικονομία. Αυτό έχει προτερήματα, αλλά έχουμε ελέγξει τα μειονεκτήματα. Υπάρχουν πολλοί θεμελιώδεις αλλαγές στη ζωή μας και όλες αυτές γίνονται εκ παραλίλου και ταχύτατα και πρέπει να εξηγήσουμε λοιπόν στους συμπολίτε μας. Πρέπει να πούμε στους συμπολίτε μας ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Γιατί μόνο ε, αν καταλάβουν οι συμπολίτε μας, αν υπάρχει διαφάνεια σε αυτές τις αλλαγές, μόνο τότε θα επιτύχουμε τη διατήρηση του τρόπου ζωής μας, την διατήρηση των αξιών μας, των συνηθιών μας, ούτως ώστε να διατηρηθεί η ιδιομορφία της Ευρώπης. Και κάτι επίσης πρέπει να είναι σαφές. Όποιο εμένει στι υπάρχουσε δομέ, όποιο δεν είναι έτοιμο να υποδεχθεί τι αλλαγέ, θα χάσει. Α ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή Ευρώπη. Εκεί που εφαρμόστηκαν θαραλέ πολιτικέ, θαραλέ μεταρρυθμίσει, εκεί πάνε καλύτερα τα πράγματα για όλου. Εκεί υπάρχουν μελλοντικέ προοπτικέ. Αυτό το διαπιστώνουμε καλύτερα στι χώρε τη κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Από που κατέρευσε ο απολυταρχικό κομμουνισμός, έγιναν τεράστιες ε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Οι πολίτες των κρατών αυτών ξέρουν καλύτερα από εμά ε, στην ε, Δύση και στον Νότο ότι το να παραμένουμε ακίνητοι η αδράνεια σημαίνει υποχώρηση. Όποιος λοιπόν εμένει στο παρελθόν δεν επιτυχάνει τίποτα. Χρειαζόμαστε ετοιμότητα για μεταρρυθμίσεις. Ας επιτρέψουμε στους πολίτες μας να είναι υπέρ της αλλαγής να είναι χαρούμενοι για τις αλλαγές. Κάτι ακόμη. Οι μεταρρυθμίσεις. Η αντικειμενικότητα. Η Ευρώπη πρέπει να είναι ρεαλιστική. Αυτό απαιτείται από κάθε χώρα μεμονωμένα. Αλλά η Ευρώπη έχει γίνει και πολύ πιο τεχνολογική. Χρησιμοποιούμε όλοι πάρα, ε, πάρα πολλά ε, μηχανήματα. Αλλά θα ήθελα να μην είμαστε μόνο τεχνοκράτες. Θα ήθελα στο μέλλον να στραφεί η Ευρώπη και προς τις ιδέες της και να γίνει πιο φιλική προς όλους. Τι εννοώ. Όταν ήμουν νέος, όταν άρχισα να ενδιαφέρομαι για την πολιτική, διάβασα πολλά για τις ευρωπαϊκές ιδέες από τους ιδρυτές της Ευρώπης. Και ε, μέσω των, εν μέσω των ερηπείων του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου υπήρξαν ιδεαλιστές που είπαν ότι θέλω μια Ευρώπη που να είναι ανοιχτή, θέλω μια Ευρώπη που να ξεπεράσει την απολυταρχία και τους εθνικισμούς, μια Ευρώπη που να επανέλθει στις ιστορικές της ρίζες. Θέλω επίσης είπαν μια Ευρώπη χωρίς ελέγχου στα σύνορα, με μια κοινή αγορά, με μια πολυμορφία, ανθρώπων που να συνεργάζονται. Αυτά μέσα στα ερήπια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μια ολόκληρη γενιά πολιτικών, δεξιών και αριστερών. Σκέφτηκαν τότε και ονειρεύτηκαν το αδιανόητο. Σήμερα μπορεί να πει κανεί, μα τι επιρμένοι ήταν. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το αδιανόητο το επέτυχαν, ενίκησαν. Και σήμερα, σήμερα συζητάμε για six pack, μιλάμε για οδηγία μη μη-feed, για μεταρρύθμιση του γεωργικού τομέα. Όλα αυτά είναι σημαντικά βεβαίω. Αλλά αρκούν. Έχει τόσο πολλά περισσότερα να προσφέρει η Ευρώπη. Η Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα. Η Μεγάλη Βρετανία είναι η γενέτειρα του κοινοβουλευτισμού. Αυτή μας εχάρισε αυτές τις ιδέες. Και σήμερα ολόκληρη η Ευρώπη είναι περήφανη για την κοινοβουλευτική της παράδοση. Η Γαλλία, η Γαλλία που χθες ήταν η εθνική της ορτή, μας ε, ε, ε, εμψύχωσε με τις ιδέες ε, της ισότητας, της ελευθερίας και της αδελφότητας για τις ισότητας ανδρών και γυναικών. Στη Γαλλία γεννήθηκαν όλες αυτές οι αρχές τις οποίες μας χάρισε σε όλους την Ευρώπη και είμαστε περήφανοι για την χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Γερμανία υπήρξε ο προτεσταντισμός η Ελλάδα με τη φιλοσοφία μας χάρισε επίσης τη φιλοσοφία και το δίκαιο και χωρίς την Ελλάδα δεν θα ήταν ε, σήμερα δυνατή η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και επίσης η Ισπανία και η Πορτογαλία μας άνοιξαν προς τον κόσμο ολόκληρο. Όλοι αυτοί λοιπόν προσέφεραν και όλοι αυτοί συνεχίζουν να προσφέρουν πολλά στην Ευρώπη. Αυτές οι κατακτήσεις είναι σήμερα τμήμα της κοινή μας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Όλοι οι Ευρωπαίοι συνέβαλαν. Όλοι οι Ευρωπαίοι ωφελήθηκαν από τους άλλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντίληψή μου για την Ευρώπη βασίζεται ακριβώς σε αυτές τις κατακτήσεις. Βεβαίως είμαστε υπέρ ε, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διαχωρισμού ε, κράτους και θρησκείας. Αλλά αυτά δεν είναι αυτονόητα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όταν ε, συναντιέται το G20 συζητάμε για θέματα εμπόριο. Αλλά ποιο λέει βεβαίως εμπόριο. Αλλά πρέπει να απαγορεύεται η παιδική εργασία. Το κάνουν αυτό στην Ινδία και τη Βραζιλία. Όχι. Εμεί οι Ευρωπαίοι πρέπει να το επιβάλλουμε αυτό. Ποιο ε, θέτει το θέμα τη καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή το κάνει αυτό η Κίνα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, όχι εμεί πρέπει να λάβουμε πρωτοβουλία. Ποιο υπενθυμίζει σε αυτές τις μεγάλες συναντήσει στον κόσμο ότι πρέπει να επιδιώκουμε να επιλύουμε και να προλαμβάνουμε τι συγκρούσει. Οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι το κάνουν αυτό. Όχι, εμεί πρέπει να τα θέσουμε αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η επιθυμία μου για τη νέα γενιά σήμερα. Μια Ευρώπη που να είναι περήφανη για την μεγάλη ιστορική της κληρονομιά πνευματική της κληρονομιά που θα σταματήσει να τσακώνεται μεταξύ της και θα παίξει το ρόλο στον κόσμο που ενσωματώνει όλες αυτές τις αρχές και τα κοινά μας στοιχεία. Εάν προωθήσουμε αυτές τις ιδέες, οι Ευρωπαίοι θα εξακολουθήσουν και θα ξαναποκτήσουν ενθουσιασμό για την Ευρώπη, περηφάνεια για την Ευρώπη, περηφάνε για το έθνος τους, αλλά συνείδηση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι έχουμε συμβάλει σε μια ανάπτυξη του πλανήτη να μην ξεχάσει η Ευρώπη τα καθήκοντά της. Γιατί ο κόσμος χρειάζεται την Ευρώπη. Ο πλανήτης χρειάζεται την Ευρώπη. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ευρώπη, πέρα από, το, από τα καθήκοντά τους, δεν θα μπορούσε να είναι και κάτι που το αγαπάμε. Η Ευρώπη με τον πολιτισμό της, με τα μνημεία της, Ξέρετε πολύ καλά ότι από όλε τι γωνιέ τη γη έρχονται στα μουσεία μα, στι ιστορικέ μα πόλει για να δουν τον πλούτο μα αυτό. Που πουθενά δεν υπάρχει τόσο πολιτιστικό πλούτο. Η Ευρώπη είναι τόσο ζωντανή, τόσο πλούσια και εγώ ω Βαβαρό, ω Γερμανό αισθάνομαι Ευρωπαίο και αισθάνομαι θαυμάσια στην Ήπειρό μου. Χαίρομαι που είμαι Ευρωπαίο. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτή η συναισθηματική πλευρά να καταστεί σαφή στους συμπολίτες μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ανασκουμποθούμε, ας εργαστούμε. Σήμερα ας δώσουμε ισχυρή εντολή στον Ζαν Κλοντ Ιούγκερ, ούτως ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Μαζί του, μαζί του εμείς ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει τη δουλειά της και απλά να τα καταφέρει. Και πιστεύω ότι πέρα από την καθημερινότητα πρέπει να έχουμε και τις γενικότερες ιδέες όπως τις είχαν οι ιδρυτές. Ιδέες που, είναι, που να είναι μια προπτική μέλλοντος για μια Ευρώπη που να είναι περήφανη για την πολυμορφία της, για τα έθνη της, αλλά επίσης ευγνώμων που είναι και έχει η Ευρωπαϊκή Συνείδηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βίβα. Για την ε, ομάδα των Σελστών και Δημοκρατών, ο κύριος Πιτέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Ιούνκερ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου μιλώντας για μια περιφέρεια που δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία όμως τα τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες έχει πραγματικά γίνει κομμάτι της Ευρώπης, τη λωρίδα της Γάζας. Υπάρχει πόλεμος εκεί. Δεν ξέρω κι εγώ στη σειρά ποιος πόλεμος είναι που κάνει χιλιάδες θύματα, που προκαλεί χιλιάδες θύματα, αμάχους. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, δεν μπορούμε να αποστρέφουμε την κεφαλή είναι κάτι που συμβαίνει στα σύνορα της Ευρώπης. Θυμηθείτε τι γίνεται στη Συρία, λίγα χιλιόμετρα από την Κύπρο. Σκεφτείτε τι γίνεται στο νότο της Ιταλίας, στη Λιβύη, στη Λωρίδα της Γάζας, στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία. Πόλεμος λοιπόν, ο πόλεμος νομίζαμε ότι τον είχαμε εξορκίσει. Επέστρεψε ο πόλεμος όμως, ξύπνησε τους παλαιούς δαίμονες. Θυμηθείτε τη Σρεμπρένιτσα, ξέρουμε ότι έχουν περάσει ε, πολλά χρόνια αλλά ενθυμούμεθα το τι συνέβη. Είναι ο καθρέφτης τον οποίο πρέπει να κοιταχτούμε για να νιώσουμε το πραγματικό νόημα της ιστορίας. και ταυτόχρονα να κατανοήσουμε την αιτία ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά είναι οικονομική και νομισματική ένωση και τραπεζική, πιστοτική ένωση. Είναι όμως και κάτι παραπάνω. Είναι ένα σχέδιο εκπολιτισμού, ειρήνης, αλληλεγγύης. Πρώτος στόχος αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου είναι πραγματικά να προσπαθήσουμε για να επιβάλλουμε την κατάπαυση του πυρός και ένα ανθρωπιστικό πρόγραμμα για τη Γάζα. Η Γάζα θα δείξει πόσο ικανή είναι η Ευρώπη. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αδρανείς μπροστά στα θύματα. Εδώ και πέντε χρόνια λοιπόν κύριε Πρόεδρε ήταν μπροστά μας ο, ο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόσο. Η κρίση είχε μόλις ξεσπάσει και πολλοί είχαν αρχίσει να προαναγγέλουν το τέλος της Ευρώπης. Πέντε χρόνια μετά και το θυμήσατε αυτό με κάθε ειλικρίνεια, η κρίση είναι μαζί μας. Η Ευρώπη πραγματικά χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη αντίδραση, υπάρχει κίνδυνο στον τομέα της απασχόλησης, υπάρχει φτώχεια. Μια ολόκληρη γενιά έχασε την ελπίδα της για το μέλλον. Ε, πολύ συχνά κύριε Γιούνκερ, πρόεδρε Γιούνκερ, γιατί πραγματίστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα μορφωμένος και αναφέρεστε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είναι σημαντική ιστορία και πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος, από τα λάθη τα οποία μας οδήγησαν στη σημερινή κρίση. Το πρώτο λάθος είναι παλαιότατο. Είναι θα έλεγα αυτό που οδήγησε και στην κρίση της δεκαετίας του 30. Λιτότητα όταν υπάρχει κρίση στη ζήτηση έπρεπε να βοηθήσουμε να ανακάμψει η παραγωγή. Έπρεπε εμείς ε, να μεταρρυθμίσουμε ε, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και όμως, στο όνομα μιας λογικής, αυστηρά λογιστικής, μειώσαμε τις επενδύσεις, μειώσαμε την κοινωνική δαπάνη. υπήρξε μια νέα σχεδίαση στον τρόπο ανάπτυξης των οικονομιών μας. Κανένας δεν θέλει φυσικά χωρίς έλεγχο να αρχίσει να αυξάνεται πάλι το δημόσιο χρέος. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εξυγίανση των δημοσιονομικών και την στήριξη σε επενδύσεις οι οποίες να βλέπουν μακριά θα πρέπει εμείς, ε, ε, κανένας δεν θα πρέπει να μην θέλει να εξηγιανθούν τα δημοσιονομικά. Αλλά ε, πώς θα το κάνουμε αυτό όταν ένας στους δύο νέους είναι άνεργος. Πού είναι η τάξη στα οικονομικά όταν η φτώχεια αυξάνεται συνέχεια. Είναι πιο σημαντική η τάξη στην κοινωνία ή η τάξη στα δημοσιονομικά. Το μεγάλο μάθημα λοιπόν αυτής της κρίσης είναι ότι οι κανόνες, το είπατε και εσείς στην παρουσίασή σας κύριε Γιούνκερ, οι κανόνες, όλοι οι κανόνες, ακόμα και οι δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να υπόκεινται στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Το δεύτερο μάθημα είναι ότι στην Ευρώπη όλοι εξαρτώμεθα από τους άλλους. Οι οικονομίες μας συνδέονται μεταξύ τους. Οι, διαταράξεις, οι αναταράξεις στις νομισματικές αγορές ε, μεταφέρονται και στις άλλες αγορές. Οι μετανάστες της Λαμπεντούζα θα περιθωριοποιηθούν σε λίγα χρόνια στις πρωτεύουσες της Ευρώπης, στη Ρώμη, στη Μαδρίτη και τα Όλα αυτά δείχνουν τις ευθύνες που έχουν και απαιτούν από μας αλληλεγγύη, απαιτούν από μας δράση και να συμμεριστούμε τα βάρη. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε μπλακεί σε αυτή την κρίση και ας το παραδεχτούμε πρόεδρε Γιούνκερ γιατί οι δεκάδες συναντήσεις κορυφών δεν κατάφεραν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Οι αποφάσεις τους ήταν ανεπαρκείς, ήταν συγκεχημένες. Απαιτείται λοιπόν μεγαλύτερη και ισχυρότερη δημοκρατία. Γι' αυτό σας στηρίξουμε. Πώς θα σας στηρίξουμε τώρα. Πιστεύουμε ότι εσείς έχετε πάρει τα μαθήματα που έπρεπε, ιδιαίτερα σε σχέση με το αίτημα για περισσότερη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν μπροστά σε μας βλέπουμε ότι έγινε μια μικρή επανάσταση στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες για πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκλέγεται λαμβάνοντας υπόψη την ψήφο των Ευρωπαίων πολιτών, ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι ένα δείγμα ενίσχυσης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και πίσω δεν θα μας οδηγήσει αυτή η απόφαση. Υπήρξε η αιμονή αν θέλετε, η επιμονή φυσικά αυτού του κοινοβουλίου και γι' αυτό το πετύχαμε. Αν δεν είχαμε υπάρξει εμείς δεν θα μπορούσατε να γίνετε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ψήφος μας ε, ε, σήμερα το απόγευμα δεν είναι μια λευκό επιταγή. Εμένα μου άρεσαν ιδιαίτερα κύριε Πρόεδρε κάποιες αναφορές τις οποίες κάνατε στα κοινωνικά θέματα και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, την οποία υπογραμμίσατε επίσης. Είναι κάτι που ανήκει στον πολιτισμό των σοσιαλιστών, των δημοκρατών και προοδευτικών στην Ευρώπη. Εσείς δεν είστε βέβαια σοσιαλιστής και δεν ζητάμε για να σας υποστηρίξουμε, αν και ποτέ δεν θα πρέπει κανείς να προκαταλάβει το μέλλον, ε, να σας ζητήσουμε να γίνετε. Εσείς κερδίσατε τις εκλογές, όχι εμείς και γι' αυτό σωστά είστε υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τους επόμενους μήνες με την ακρόαση των υποψηφίων επιτρόπων θα επαληθεύσουμε τη συμβατότητα ανάμεσα στο δικό μας πρόγραμμα και το πρόγραμμα της Μελλοντικής Επιτροπής. Θα είμαστε απόλυτοι. Ο Δημοκρατικός Κοινοβουλευτικός Έλεγχος επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ενισχυθεί. Η συζήτηση για το καθεστώς των πραγμάτων στην Ευρώπη δεν θα είναι μια ρητορική συζήτηση, αλλά θα καταστεί μια ετήσια πραγματική αξιολόγηση της κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς δεν απλά θέλουμε να τιμήσουμε τη νέα κοινοβουλευτική δημοκρατία ίσα ίσα. Τις τελευταίες μέρες όπως γνωρίζετε διαπραγματευθήκαμε και καταθέσαμε τις προτεραιότητές μας. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Ζητήσαμε περισσότερες επενδύσεις για μεγαλύτερη ανάπτυξη, μια πιο κοινωνική Ευρώπη, περισσότερη αλληλεγγύη, ιδιαίτερα σε σχέση με τα θέματα της μετανάστευσης. Στις ερωτήσεις μας εσείς σήμερα το πρωί και στο γραπτό σας κείμενο και στην προφορική σας παρουσίαση δώσατε απαντήσεις, απαντήσεις που πείθουν. Σας ζητούσαμε συγκεκριμένους αριθμούς, συγκεκριμένα στοιχεία. Εμείς μας δώσατε κάποια στοιχεία, μας δώσατε και μια χρονική προθεσμία. Είπατε 300 δις για ένα πρόγραμμα επενδύσεων που θα δημιουργήσει πλούτο και ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Και είπατε ότι θα ξεκινήσετε το Φεβρουάριο του 2015. Εσείς εμείνατε και στο θέμα της βιομηχανικής πολιτικής, κάτι το οποίο για πάρα πολύ καιρό ε, δεν θέλαν να το αγγίξουν οι φιλελεύθεροι. Λοιπόν, αυτό θα βοηθήσει αν φτάσουμε ε, στη βιομηχανική παραγωγή να αντιπροσωπεύει το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Επίσης, καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, αναθεώρηση της οδηγίας για τις αποσπάσεις των εργαζομένων, σεβασμός της αρχής, η οποία λέει για την ίδια εργασία, ίδια αμοιβή. Ταυτόχρονα δεσπευθήκατε και για την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ μέσω της υιοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μιας κοινή βάσης φορολογικής επιβολής για τις επιχειρήσεις όπως επίσης και μια σωστή εφαρμογή ε, του φόρου για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ταυτόχρονα αντιμετώπιση των προβλημάτων χωρών όπως η Ελλάδα και όλων των άλλων χωρών που κινούνται στα πλαίσια προγραμμάτων στήριξη των μεταρρυθμιστικών εθνικών προσπαθειών, έγκριση της οδηγίας κατά των διακρίσεων η οποία δυστυχώς δεν έχει προωθηθεί λόγω των λανθασμένων αποφάσεων των, των συναντήσεων κορυφής. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βοηθήσουμε το μέγιστο αριθμό νέων να επωφεληθούν από την εγγύηση, από το Ταμείο Εγγύησης για τους νέους. Λοιπόν, πολλά έχουμε πετύχει, πολλά μένουν να πετύχουμε και γι' αυτό θα σας στηρίξουμε. Πολλά μπαίνει να γίνουν, επαναλαμβάνω. Θα θέλαμε περισσότερα από πλευρά σας για το θέμα της ευελιξίας. Εσείς περιοριστήκατε στο να μας υπενθυμίσετε τη συμβουλία του Συμβουλίου πάνω σε αυτό. Εμείς ζητήσαμε περισσότερα στοιχεία για τον προσανατολισμό, για ε, για το διορισμό του Επιτρόπου του Υπεύθυνου για το ΕΚΟΦΗΝ ε, ενός στελέχους των σοσιαλιστών. Δεν έχουμε απαντήσεις εδώ, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να στηρίξουμε τις χώρες οι οποίες κάνουν μεταρρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει οι χώρες αυτές να μην ε, αντιμετωπίσουν περισσότερα προβλήματα λόγω κάποιων επιβαλόμενων εκ των έξω δημοσιονομικών κανόνων. Θέλουμε περισσότερα για την ανάπτυξη, θέλουμε περισσότερα στοιχεία για τις γονικές άδειε, γιατί θέλουμε οι γυναίκες της Ευρώπης να συνδυάσουν την επαγγελματική ζωή και την οικογενειακή ζωή. Θέλαμε να μας πείτε περισσότερα και για την περιβαλλοντική αηφορία, για το δικό μας πρότυπο ανάπτυξης, το οποίο θα πρέπει να φροντίσει το τι συμβαίνει στον πλανήτη. Θέλαμε περισσότερα στοιχεία για τη γνώση, το ταλέντο, τις ικανότητες του ανθρώπινου ευρωπαϊκού δυναμικού. Δεν θα μείνουμε αδρανείς, θα είμαστε ειλικρινεί συνομιλητές αλλά απαιτητικοί συνομιλητές. Δεν έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Αν επικρατήσει ο συντηρητισμός και η αδράνεια, σε πέντε χρόνια η Ευρώπη θα είναι μια μικρή, εξασθενημένη, φοβισμένη και διαιρεμένη Ευρώπη. Μπορούμε αντίθετα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και χάρη στις προσπάθειες όλων να ξαναθέσουμε την Ευρώπη στην υπηρεσία των πολιτών. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Ε, ξεκινάμε από διαφορετικές θέσεις, ξεκινάμε από διαφορετικές ιστορίες, αλλά τίνουμε χείρα φιλίας, χείρα εμπιστοσύνης και σας ζητάμε να μην μας προδώσετε τα επόμενα πέντε χρόνια. Θα σας παρακολουθήσουμε προσεκτικά. Καλή τύχη, Πρόεδρε Γιούνκερ. Ευχαριστώ κύριε Πιτέλα και τώρα το λόγο για την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κύριος Καμάλ. Κύριε Γιουνκερή, οι αλλαγές δεν γίνονται από μόνες τους, χρειάζονται ηγεσία. Χρειάζονται μια ηγεσία που να κοιτάζει μπροστά, όχι πίσω. Χρειάζεται μια ηγεσία που να αναγνωρίζει τις προκλήσεις του σήμερα, του 2050, όχι του 1950. Πρέπει επίσης να αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες του κόσμου που θέλει συνεργασία. Θέλει μια Ευρώπη με συνεργασία και όχι με κεντρική δίκηση. Θέλει μια ατζέντα η οποία να ανοίγει ένα όραμα μπροστά. Εμείς αυτά θέλουμε. Δεν θέλουμε μια παλιά ατζέντα. Θέλουμε οικοδομημένες νέες αναλλακτικέ λύσεις. Εσείς λοιπόν πρέπει να διευκρινίσετε τις θέσεις σας κύριε Γιούγκερ. για θέματα όπως είναι η άδεια μητρότητας, όπως είναι η δημοσιονομική λιτότητα. Εσείς είπατε και σε εμά ένα πράγμα και σε άλλες ομάδες φαίνεται ότι είπατε κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε κύριε Γιούγκερ να σηκωθείτε και να μας πείτε τι πραγματικά πιστεύετε. Όμως γνωρίζετε ότι στην πραγματικότητα, το ξέρετε και εσείς και εμείς, ότι δεν είναι αυτό που τόσο πολύ μέζει, έτσι, που νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς η ζημιά έχει γίνει. Οι εκλογές τελικά οδήγησαν σε συνεννοήσεις πίσω στους διαδρόμους. Ξέρετε κι εσείς, όπως ξέρουμε κι εμείς, ότι θα είσαστε κατά πάσα πιθανότητα ο νέο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κύριε Γιούνκερ, εμεί σα ευχόμαστε ότι καλύτερο. Αλλά τα μέλη τη δικιά μου πολιτική ομάδα δεν θα μπορέσουν να σα ψηφίσουν σήμερα για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί εμείς δεν συμφωνούμε με την διαδικασία η οποία σας οδήγησε εδώ. Δεν πιστεύουμε ότι εσείς έχετε εντολή ευρεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση από όλες τις χώρες μέλη. Και δεύτερον, γιατί τα μέλη της ομάδας μου δεν είναι πεπισμένα ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσετε μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ελπίζω τα επόμενα χρόνια να αποδείξετε ότι έχουμε άδικο. Αλλά εσεί έχετε τι προκλήσει μπροστά σα. Θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι η τελευταία του παλιού, παλιό, των παλιών συνηθιών και η πρώτη νέα. Εμείς θέλουμε μια ηγεσία η οποία θα κάνει μεταρρυθμίσεις στον προπολογισμό. Θέλουμε να ε, βγούμε μακριά από αυτή την ιδέα που λέει όσο πιο πολλά χρήματα έχουμε τόσο καλύτερο. Όχι, εμείς θέλουμε ένα καλύτερο προπολογισμό, να επενδύει, να διευκολύνει τις επενδύσεις σε υποδομές, σε τεχνολογία, σε έρευνα. Τα παιδιά μας ε, θέλουμε να κληρονομήσουν μια καλή οικονομία για το μέλλον. Δεν θέλουμε να κληρονομήσουν χρέη τα οποία χτίστηκαν κατά το παρελθόν. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε να δούμε πώ θα βρούμε περισσότερα χρήματα από του ίδιου πόρου μα, α κάνουμε μια άλλη συζήτηση. Να δούμε πώ θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα χρήματα των φορολογούμενων. Και γι' αυτό η ομάδα μου θέλει μια αφοσιωμένη επιτροπή, αφοσιωμένη στον έλεγχο του προπολογισμού. Θέλουμε ηγεσία για να έχουμε την ενιαία αγορά, η οποία να είναι κατάλληλη για, την, για το μέλλον. Θέλουμε υπηρεσίε και ενιαία αγορά που όμω δυστυχώ βρίσκονται ακόμα μακριά από την πραγματικότητα. Γιατί δεν καθόμαστε κάτω με του επιχειρηματίε και να ρωτήσουμε του επιχειρηματίε τι φραγμού συναντάνε μπροστά τι δυσκολίες έχουν. Μα ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να φέρουμε αποτελέσματα σε αυτήν την ενιαία αγορά για όλους. Ενεργειακή επίσης αγορά και εδώ πρέπει να έρθουν οι φραγμοί. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα στους καταναλωτές για ενεργειακή επάρκεια, επενδύσεις για την ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια. Θέλουμε επίσης περισσότερα δίκτυα για να έχουμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία από την Μέση Ανατολή και την Ρωσία στον ενεργειακό τομέα. Επίσης θέλουμε κίνητρα υπέρ του εμπορίου, νέες πολιτικές κατάλληλες για μια νέα εποχή. Επίσης θέλουμε περισσότερη διαφάνεια στις συμφωνίες που γίνονται με τις αναδυόμενες οικονομίες. Θέλουμε όμως και διεθνή προγράμματα για το copyright, για νέα συστήματα νομικής δικαιοσύνης. Θέλουμε η, επίσης απασχόληση σε τοπικό επίπεδο. Θέλουμε μια ηγεσία για να προωθήσει καλύτερη ρύθμιση για αυτή τη νέα εποχή στην οποία μπαίνουμε. Δεν θέλουμε κάτι το οποίο να ταιριάσει σε όλα. Θέλουμε να δούμε τι χρειάζεται για περισσότερη απασχόληση κάθε φορά. Και θέλουμε ηγεσία για να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν στην Ευρωζώνη. Τα προβλήματα με την ανταγωνιστικότητα, με την ανεργία, τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Νότια Ευρώπη. Πολλές χώρες έχουν ε, αδυναμίες και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα και είδαμε να περνάνε τα βάρη των τραπεζών, τα χρέη των τραπεζών στους φορολογούμενους τα κράτη να παρεμβαίνουν. Εμείς θέλουμε ηγεσία επίσης σε θέματα μετανάστευσης, να νιώθουν ασφαλείς οι άνθρωποι, να μπορούν να διακινούνται ελεύθερα οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να εργάζονται και να συνεισφέρουν σε νέες χώρες, αλλά να ελέγχουμε τη μετανάστευση για να γίνονται σεβαστά ε, τα δικαιώματα όλων των χωρών μελών και να φροντίσουμε και για τις χώρες εκείνες οι οποίες χάνουν τους νέους ταλαντούχους τους οι οποίοι μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Σήμερα άκουσα διάφορα παραδείγματα, μάλλον ακούσατε παραδείγματα από μένα για το που χρειάζεται ηγεσία για να μπούμε σε αυτή τη νέα εποχή, για να μην βρεθούμε στον προηγούμενο αιώνα. Θέλουμε ηγεσία για να αντιμετωπιστούν οι υποψίες και ανησυχίε των ε, πολιτών μας, για να επιβεβαιωθούν οι ελπίδες των νέων. Χρειάζεται ηγεσία κύριε Γιούγκερ. Πολλοί από τους ευρωβουλευτές της ομάδας μου δεν θα σας υπερψηφίσουν σήμερα γιατί ανησυχούν ότι δεν υπάρχει αυτή η ηγεσία. Θέλουμε όμως και ελπίζω εσείς να καταφέρετε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις αυτές και στο μέλλον να κερδίσετε έτσι την εμπιστοσύνη μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καμάλ. Για τους φιλελεύθερους τώρα, Άλντε, ο κύριος Φερχόφστατ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι ιστορική μέρα σήμερα, όχι λόγω όλων των ε, μεγαλοστομιών που ακούσαμε σήμερα το πρωί, αλλά γιατί θα εκλέξουμε έναν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με διαφορετικό τρόπο, όχι απλώς επικυρώνοντας ε, την επιλογή του Συμβουλίου, αλλά συμμετέχοντας στον καθορισμό του υποψηφίου. Και κυρίως ε, επειδή οι εκλογείς είχαν τον αποφασιστικό λόγο. Υπερψηφίζοντας σήμερα τον κύριο Γιόνκερ, ας το πούμε ανοιχτά. Καταλαβαίνω ότι ένα τμήμα του σώματος ε, δύσκολα θα το αποδεχθεί, αλλά ας το πούμε. Επιλέγοντας και εκλέγοντας ε, τον κύριο Γιούνκερ σήμερα, δημιουργούμε μια για πάντα ουσιώδη, πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατία, όπου οι πολίτες αποφασίζουν. Συνάδελφοι, δεν είναι τυχαίο είναι αποτέλεσμα μιας μακράς, ιδιαίτερα μακράς πορείας. Λόγω της ε, συμβατικής συνέλευσης, ε, συντακτικής συνέλευσης που δημιουργήσαμε το 2001 και λόγω της επιμονής κάποιων κοινοβουλευτικών. Τουλάχιστον δύο αφοσιωμένων Ευρωπαίων που θέλω να αναφέρω. Τον Άντρου Νταφ και τον Έλμαρ Μπροκ. Ο Άντρου που δεν είναι πλέον ε, συνάδελφος και ο Έλμαρ που κατά τη γνώμη μου θα εξακολουθήσει αενάως να είναι παρόν. Αλλά ναι βέβαια αυτή τη στιγμή είναι απόν, ενώ συνήθω είναι εδώ, στη θέση 263. Εξακολουθούν να φιλονικούν για το ποιος επινόησε αυτή την πρόταση στη συντακτική συνέλευση για να εκλέγεται έτσι με αυτή τη διαδικασία που σήμερα ολοκληρώνουμε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ζαν Κλοντ δεν είναι λοιπόν θέμα ότι εκλέγουμε εσένα. Πρέπει να σου το πω μήνυμα, το μήνυμα σήμερα αφορά τους συναδέλφους της, στις μεγάλες πολιτικές ομάδες κυρίως που θέλουν να σε καταψηφίσουν. Θέλω να πω στους συναδέλφους αυτές τις δύο μεγάλες πολιτικές ομάδες και και από τις άλλες ότι καταψηφίζοντας τον κύριο Γιούγκερ τι κάνουν συντάσσονται με τους ε, αντιευρωπαϊστές δηλαδή διαψεύδουν τις προσδοκίες των ψηφοφόρων τους, οι οποίοι ζήτησαν ακριβώς η δική τους επιλογή να γίνει σεβαστή και η επιλογή τους ήταν ο κύριος Γιούνκερ. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα αντιφατικό αυτό. Υπάρχουν βεβαίως αυτοί που είναι κατά της Ευρώπης, που θέλει να αγνοήσουμε την ε, επιβολή ε, της θέλησης των ε, ψηφοφόρων. Αυτούς λοιπόν θα ενισχύσετε. Εμείς όμως θα σας υπερψηφίσουμε. Δίνουμε ένα σαφές θετικό μήνυμα επίσης γιατί δεχθήκατε μια σειρά από τις προτάσεις μας. Κυρίως η πρότασή μας ήταν ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτή η υποχρέωση να διαλέξουμε μεταξύ Λιτότητα και ανάπτυξης. Σαν να αντιφάσκουν αυτά τα δύο. Ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να συνδυαστούν μετά από πέντε χρόνια, ελπίζω να ηγηθείτε μια επιτροπής που θα επιχειρήσει και τα δύο. Και δημοσιονομική πειθαρχία από τη μία, αλλά και ανάπτυξη από την άλλη. Όλοι ξέρουμε, χωρίς δημοσιονομική πειθαρχία, χωρίς σεβασμό του σύμφωνου σταθερότητα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Και παράλληλα, επίση γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη, Πρέπει να ξεπεράσουμε την απλή δημοσιονομική πειθαρχία. Πρέπει να έχουμε ένα πακέτο ανάπτυξης όπως το προτείνατε στο πρόγραμμά σας. Ο δεύτερος λόγος, ε, κύριε Γιούγκερ, για τον οποίο ε, χαιρόμαστε για το πρόγραμμά σας και θα σας στηρίξουμε είναι γιατί κάνατε μερικές σημαντικές επισημάνσεις επιτέλους συζητάμε για την νόμιμη μετανάστευση ήταν απαγορευμένο θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης μιλήσατε για τις αξίες και ότι θα αναθέσετε ε, σε έναν ειδικό επίτροπο την ε, φροντίδα για την τήρηση του κράτους δικαίου. Αλλά με κάτι διαφωνώ μαζί σας. Ανεξάρτητα από τις ε, πολιτιστικές καταβολές και τις κοινοβουλευτικές παραδόσεις, οι θεμελιώδεις αξίες είναι αδιαπραγμάτευτες και πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους ανεξάρτητα των παραδόσεών τους. Και η τρίτη δέσμευση που αναλάβατε πολύ σημαντική για μας είναι, είναι ότι η Επιτροπή σας θα έχει ε, ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Αυτός είναι ο στόχος σας, ελπίζω να τον επιτύχετε. Τέλος κύριε Γιούγκερ, έχω τα εξής τρία αιτήματα. Βεβαίως τώρα θα εκλεγείτε επικεφαλής ε, της Επιτροπής, οπότε θέλουμε τα εξής τρία. Πρώτον, να επανέλθουμε στην κοινοτική μέθοδο. Γιατί οι διακυβερνητικοί διακανονισμοί των τελευταίων πέντε ετών δεν ήταν παράδειγμα σωστή διακυβέρνηση. Δεύτερον και πιο σημαντικό, παρακαλώ, παρακαλώ, μην κάνετε όπω ο προκάτοχό σα. Αξιοποιήστε το δικαίωμα πρωτοβουλία. Μην αρχίσετε τώρα αυτά τα ταξιδάκια στο Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο και τη Ρώμη πριν θέσετε νομοθετήματα ενώπιον ε, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Κάντε το, να έχετε το κουράγιο να υποβάλλετε προτάσει. Και όχι επειδή υπάρχει μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και να μην ακούτε μόνο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καμιά φορά, εγώ θα προτιμούσα κάθε μέρα, να ακούτε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί είμαστε ισότιμοι νομοθέτες. Και επιτέλους δημιουργήστε μία νέα προοπτική, ένα, νέο όραμα για την Ευρώπη. Γιατί βλέπετε πόσο είναι χαμένοι πολλοί συμπολίτες μας, γιατί δεν υπάρχει όραμα ένα όρμα που να λέει ότι μόνο μέσω περισσότερης ενοποίησης θα ξεφύγουμε από την κρίση, όπως το επιτύχαμε στη δεκαετία του 80. Και αν το επιτύχετε αυτό θα μας βρείτε, εάν εργαστείτε προς αυτή την κατεύθυνση, θα είμαστε και 68 φιλελεύθεροι βουλευτές στο πλευρό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Για την ενιαία αριστερά η κυρία Τσίμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Γιούγκερ. Αντιτίθεται, αντιτίθεμε ε, όχι με, μεγάλη, με μεγάλο ενθουσιασμό, όχι επειδή είναι ο χαρακτήρας μου ε, τέτοιος σε ορισμένα που υπόθηκαν στη γενική εφορία. Το κάνω όμως γιατί δεν πιστεύω ορισμένες ε, διαπιστώσεις. Ναι βέβαιως κάναμε ένα βήμα. Μέσω των ε, εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζουμε και το ποιο θα ηγηθεί της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι αυτό. Αλλά λέω όχι εάν αυτό θεωρείται ότι είναι η τεράστια νίκη της δημοκρατίας. Όχι, είναι μόνο μια αρχή. Και είμαστε μόνο στην αρχή, γιατί αυτό το μικρό πρώτο βήμα αξιοποιήθηκε ελάχιστα τις τελευταίες εβδομάδες, τους περασμένους μήνες, ούτως ώστε να υπάρξει μια αξιόπιστη δημοκρατική πρόοδος για την Ένωση. Υπόθηκε ότι είναι κατάκτηση και ότι παράλληλα διαπιστώνουμε ότι υπήρξε ένα παζάρι για τη διανομή αξιωμάτων όπου βλέπουμε ότι οι μεγάλοι συνασπισμοί κυριαρχούν Κατά τη γνώμη μου, αυτό όμως είναι αποτυχία της δημοκρατίας, για την οποία μίλησε ο κύριος Χάμπεμας. Βεβαίως δεν είναι κατάρρευση. Πρέπει όμως να αναπτύξουμε περισσότερο την ε, δημοκρατία, να δούμε το αποτέλεσμα των εκλογών καλύτερα. Δεν ισχύει ότι κέρδισαν οι συντηρητικοί. Σχεδόν 3,5 φορές από τις ψήφους των συντηρητικών ψήφισαν αλλιώ. και αναφέρομαι σε εκείνους που απήχων ή σε εκείνους ή για εκείνους που θεωρούν ότι λόγω των επιπτώσεων που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια δεν θέλουν κανένα μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουν να επανέλθουν σε εθνικές απαντήσεις, σε εθνικές διεκδικήσεις. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο κατά τη γνώμη μου και τροποποιεί τη δημοκρατία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι χάσαμε αυτές τις εκλογές. Συγκεκριμένα όλοι εκείνοι που θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια ένωση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης. Όλοι αυτοί που θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι δύναμη ειρήνης, να παίξει ένα διαφορετικό ρόλο για την εξωτερική πολιτική. Αυτό που ήταν η αρχική προοπτική, το αρχικό όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο κοντά και όχι να τους απομακρύνει. Και τα τελευταία χρόνια συνέβη το αντίθετο. Γι' αυτό όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι τόσο ικανοποιημένοι και τόσο χαρούμενοι να κάνουν ό,τι πρέπει ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα όραμα για το μέλλον για όλους τους πολίτες. Το μήνυμα που διαπιστώσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, τους μήνες, τα χρόνια ήταν ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Καμία εναλλακτική λύση στην πολιτική της ριζοσπαστικής επικράτησης των αγορών, της στήριξης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της καταστροφής του κοινωνικού προτύπου, των ιδιωτικοποιήσεων των δημοσίων υπηρεσιών, της φιλελευθεροποίησης, απορρίθμισης των ε, συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικών προδιαγραφών. Προς το συμφέρον της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οργανωμένης οικονομίας και των χρηματαγορών. Αυτά είναι μια επανάληψη αυτών που έλεγε η παλιά Βρετανή Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει άλλη ανακτική λύση. Και όλοι όσοι έχουν άλλη άποψη αντιμετωπίζουν ένα τείχο και έχουν απομακρυνθεί όλο και περισσότερο από την Ένωση. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζετε και εσείς κύριε Γιούνκερ και όλοι μα. και για την οποία νομίζουμε ότι πρέπει να εξαγάγεται διδάγματα από τις εκλογές. Υπάρχει μια τεράστια ρήξη στην ευρωπαϊκή πολιτική. Η εικόνα που μας δώσατε είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως στο παρελθόν. Θα συνεχίσουμε ό,τι κάναμε και στο παρελθόν. Αυτό δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Από εσά αναμένουμε σαφείς απαντήσεις για το πώς πρέπει να αλλάξει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τρόικα. Δεν μας ικανοποιεί το ότι λέτε ότι η Τρόικα πρέπει να γίνει πιο δημοκρατική. Μα τι σημαίνει αυτό. Μέσω της συμμετοχής κάποιων κοινοβουλίων. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η πολιτική της Τρόικας που στην ουσία επηρεάζει τη συνταγματική τάξη των χωρών προσαρμογής. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Καταστρέφει τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το καθήκον. Τι θα προτείνετε εναλλακτικά. Δεν αρκεί απλώς να λέτε να φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι απαντήσεις έχετε εσείς. Ιδιαίτερα ε, λόγω και του ρόλου της Κομισιόν στην Τρόικα για τα χρέη, για το πώς θα αντιμετωπιστεί το χρέος, για το πώς θα υπάρξουν μειώσεις των χρεών. Πώς θα το κάνετε αυτό. Είπατε ότι θα υπάρχουν και πολλά κοινωνικά θέματα στο κέντρο των προσπαθειών σας. Βεβαίως, μας ικανοποιεί αυτό. Αλλά πολύ συχνά έχουμε ακούσει παρόμοιες δηλώσεις τα τελευταία χρόνια. Τα ίδια και τα ίδια. Θέλουμε συγκεκριμένα να μας πείτε. Πώς θα το επιτύχετε αυτό. Αναφερθήκατε σε ελάχιστες αποδοχές στα κράτη-μέλη. Σημαντικό. Αλλά αυτό, αυτός ο ελάχιστος μισθός, οι ελάχιστες αποδοχές θα επαρκούν για να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας. Τα επιδόματα θα επαρκούν. Αυτό είναι το αποφασιστικό. Και καταλήγω. Κάτι ακόμη. Ήρθατε στην ομάδα μας, απαντήσατε ερωτήσεις ή σε ορισμένες δεν απαντήσατε. Αλλά αυτό που πάντα τονίσαμε είναι ότι αναμένουμε από εσάς ως Προέδρου της Κομισιόν για τα μεγάλα προβλήματα εντός της Ένωσης να είστε πολύ πιο αποφασιστικός. Για παράδειγμα, η κατάσταση στην Κύπρο. Ποιος αν όχι εσείς δεν θα έπρεπε να στραφείτε προς την Τουρκία. Και αναμένω και για την ε, Ουκρανία. Είπατε επίσης ότι για τη Ρωσία δεν θα, δεν θα επιτρέψετε οι, όλοι να κατηγορούν τη Ρωσία για όλα. Θέλουμε μια Ευρώπη που να τους ε, ε, περιλαμβάνει όλους, που να μην προκαλέσει νέες διχόνοιες. Δεν θα σας υπερψηφίσουμε σήμερα κύριε Γιούγκερ, αλλά την καθημερινή δραστηριότητά σας θα την παρατηρούμε και όπου προτείνετε βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων θα σε υποστηρίξουμε. Για τους πρασίνους, ο κύριος Λαμπέα. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν έχουμε 27 εκατομμύρια ανέργων και 25% των νέων είναι χωρίς ε, προοπτικές για το μέλλον, 25% είναι στα όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού. Όταν 10% από εμά τους Ευρωπαίους κατέχουμε το 60% του συλλογικού πλούτου των Ευρωπαίων, σημαίνει ότι κινδυνεύουν οι κοινωνίες μας όταν ε, έχουμε απορρίθμιση στα θέματα του κλίματος, όταν δεν μπορούμε να μειώσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας, όταν οι ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας έχουν κατανοηθεί με τέτοιο τρόπο τον, ε, οι μη ανανεώσιμε έχουν κατανοηθεί με τέτοιο τρόπο τα τελευταία χρόνια, η ίδια η ύπαρξη των κοινωνιών μας απειλείται. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, οι κυβερνήσεις που εκλέγονται δημοκρατικά υφίστανται καθημερινή απειλή και εκβιασμούς από τις οικονομικές αγορές, από τα δημοσιονομικά ιδρύματα που λένε ότι είναι πολύ μεγάλα για να αποτύχουν, όταν έχουμε όλο και περισσότερους ειδικού αξιωματούχους που δεν εκλέγονται και όταν ε, στο όνομα της ελευθερίας ή και του κέρδους ακόμα ιδιωτική μας ζωή και ελευθερία αμφισβητείται, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η δημοκρατία. Αγαπητοί φίλοι, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Συνεπώς, κύριε Γιούγκερ, είσαστε εσείς ο άνθρωπος για μια πραγματική δημοσιονομική ένωση, γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν βιώσιμα δημοσιονομικά χωρίς να υπάρχει έλεγχος των δαπανών, αλλά και βιώσιμα έσοδα. Όταν λοιπόν τόσα χρήματα κάθε χρόνο όταν ε, δεν υπάρχει διαφάνεια και υπάρχει αντίθετα νομιμοποίηση του παράνομου χρήματος, τότε βέβαια κινδυνεύει αυτή η Δημοσιονομική Ένωση. Δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον για ένα ενιαίο νόμισμα χωρίς δημοσιονομική αλληλεγγύη μέσα σε μια οικονομική ζώνη. Κύριε Γιούνκερ, είσαστε εσεί ο άνθρωπος για μια κοινωνική ένωση η οποία να αντικαταστήσει το δόγμα του ανταγωνισμού ανάμεσα στα συστήματα κοινωνικής μας προστασίας και που θα προσφέρει σύγκληση των συστημάτων αυτών. Θα φροντίσετε να υπάρχει ένας ελάχιστος μισθός, ελάχιστα έσοδα και ε, θα σταματήσετε αυτή την πρωτοβουλία που ονομάζεται Ρίφιρ και που πολλοί στερίζουν εδώ πέρα που τελικά καταλήγει στην μείωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας προδιαγραφών όπως γίνεται στην Αμερική. Θα είσαστε εσείς ο άνθρωπος της Ενεργειακής Ένωσης που δεν θα είναι απλώς ένα συνδικάτο αγοράς ε, φυσικού αερίου αλλά θα αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο ενεργειακής πολιτικής που με τις ανανεώσιμες πηγές, με την ενεργειακή απόδοση, με δίκτυα διανομής ενέργειας θα καταστήσει την Ευρώπη πρωταθλητή στον κόσμο για την οικολογική αλλαγή στην οικονομία μας. Θα είσαστε εσείς ο άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει η Ευρώπη να εκφράζεται με μία φωνή και που δεν θα υφίσταται απλώς τις αποφάσεις του Πούτιν όπως έγινε στην Ουκρανία ή και σε άλλες περιπτώσεις αν λάβουμε υπόψη μας στην Μέση Ανατολή και όλες τις ε, Συγκρούσει που έχουμε εκεί. Και θα τελειώσω και με κάτι άλλο. Κύριε Γιούνκερ, θα είσαστε εσείς ο άνθρωπο τη επαναδημοκρατικοποίηση, όχι μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τη Ευρώπη ολόκληρη. Γιατί σήμερα αυτό είναι που ενδιαφέρει του συμπολίτε μα. όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια πρέπει να εμπλέκονται στις πολιτικές αποφάσεις. Είσαστε εσείς ο κατάλληλος άνθρωπος, ώστε οι αποφάσεις να εφαρμόζονται όταν πρόκειται για θέματα που τους ε, αφορούν. Είσαι στο κατάλληλο άνθρωπο που θα φροντίσει οι συμπολίτε μα να εμπλέκονται άμεσα. Έχουμε ευτυχώ την πρωτοβουλία των πολιτών. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πιο συμμετοχική δημοκρατία. Τα λόμπι, όποιοι είδου και να είναι, να κοιτάνε τη δικιά του τη δουλειά και δεν είναι δικιά τους δουλειά να γράφουν τους νόμους της Ευρώπης. Σας άκουσα λοιπόν και θα μπορούσα να σας πιστέψω. Σας έχω γνωρίσει και από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, το ξέρετε, δεν έχουμε πάντα τις ίδιες απόψεις, αλλά έχουμε την τάση να σας πιστέψουμε. Συγχρόνως όμως ε, δυσπιστούμε, γιατί ποιοι είναι αυτοί που σας στηρίζουν σήμερα. Οι τρεις κύριες πολιτικές οικογένειες που σας στηρίζουν ε, σήμερα είναι ακριβώς αυτές οι οικογένειες που είναι στην εξουσία στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Αν θέλανε να έχουν αλλάξει κάτι θα το είχαν ήδη κάνει, έτσι δεν είναι. Εξάλλου, δεν μπορώ να θυμηθώ και αυτό που άκουσα χτες στον ε, κύριο Τράγκη στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για διαρθρωτικές αλλαγές, για μείωση των δαπανών, μείωση της φορολογίας, αύξηση της ελαστικότητας στην εργασία για αυτόν. Ό,τι έγινε στις 25 Μαΐου δεν μετράει καθόλου από ό,τι φαίνεται. Και τέλος θα σας πω και το εξή. Είμαστε μοιρασμένοι στην ομάδα μου, γιατί πολλοί στηρίζουμε βέβαια το μηχανισμό που σας οδήγησε μέχρι εδώ, αυτή τη διαδικασία, που είναι βέβαια ένα μικρό βήμα, αλλά πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό. Δεν θα φτάσουμε βέβαια σε δημοκρατική επανάσταση από αυτό και μόνο, αλλά θέλουμε η Ευρώπη να γίνει ένα πιο δημοκρατικό όργανο. Οπότε είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, γι' αυτό και πολλοί από εμά θα σας στηρίξουν. Όμως, μια άλλη, ε, κάποια άλλη στην ομάδα δεν έχουν εμπιστοσύνη, γιατί βλέπουν ποιοι σας στηρίζουν σήμερα και αναρωτιούνται θα μπορέσετε να κάνετε αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη. Όποιο πάντως και αν είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κύριε Γιούγκερ να ξέρετε ότι κάθε φορά που η Επιτροπή σας εδώ στο σώμα θα προτείνει προτάσεις οι οποίες είναι τολμηρές και θα φροντίσουν ο χώρος αυτός της Ευρώπης να γίνει χώρος βιώσιμης ευημερίας για όλους και πανίδρες της δημοκρατίας, τότε να ξέρετε ότι θα έχετε την ομάδα μας στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λαμπέα για την ε, Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας ο κύριος Φάραντς, η FDD. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Αν αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία στην πραγματικότητα, να το ξανασκεφτούμε θα πρότεινα. Μα είπατε ότι λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών ο κύριο Γιούνκερ ε, εδώ παρόν ε, είναι ο υποψήφιο που πρέπει να εγκρίνουμε. Αλλά κανένα στο Ευρωπαϊκό δεν τον γνώριζε όταν ψηφίζανε τι ευρωεκλογέ δεν ήξεραν ότι σχετίζεται με τον επόμενο πρόεδρο της Επιτροπής και οι ψηφοφόροι σας και στις δικές σας χώρες δεν κατάλαβαν περί σε πρόκειται. Το όνομα του κυρίου Γιούγκερ δεν ήταν σε κανένα ψηφοδέλτιο, σε καμία χώρα. Και όλη αυτή η διαδικασία ήταν πραγματικά απίστευτη μηχανογραφία. Διότι αυτός που έχασε ο κύριος Σούλτ παίρνει ως βραβείο παρηγοριά πρωτοφανή δεύτερη θητεία Προέδρου του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά είναι κοροϊδία αύξηση τη δημοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το εκλεγμένο τμήμα των ευρωπαϊκών θεσμών, είχε λόγο και αποφάσισε αν ο κύριο Γιούνκερ πρόκειτο να γίνει πρόεδρος της Επιτροπής λέγεται. Αλλά σκεφτούμε τι διαδικασία ακριβώ κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μα ζητείτε να ψηφίσουμε, αλλά υπάρχει μόνο ένα υποψήφιο. Ωραία, σαν τον παλιό καλό καιρό τη Σοβιετική Ένωση. Για μένα δημοκρατία χρειάζεται πάνω από έναν υποψήφιο, αλλά δεν είναι το χειρότερο αυτό. Καθόλου το χειρότερο. Θα είναι μυστική η ψηφοφορία. Απίστευτο. Απίστευτο. Έγιναν ε, ευρωεκλογέ, αλλά τώρα οι ψηφοφόροι, οι ψηφοφόροι μα δεν θα ξέρουν τι ψήφισε ο καθένα. Κύριε Σούλτ, είστε πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Σε εσά απευθύνομαι δεν θα πρέπει να είναι μυστική ψηφοφορία. Εφόσον είμαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι, θα πρέπει να είμαστε υπόλογοι για τι ενέργειέ μα έναντι των ψηφοφόρων μα. Και να μην υπάρχει μυστική ψηφοφορία. Αυτό είναι τεράστια προσβολή έναντι των εκλογέων. Επίσης, μετά από την τεράστια αύξηση του ποσοστού ψήφων των ευρωσκεπτικιστών, κάποιοι θα αναθεωρούσαν τι απόψει τους αλλά όχι. Ο κύριος Κάμερον έκανε μια αδύναμη προσπάθεια να αντισταθεί στο Γιούγκερ αλλά κυρίω τον απασχολούσαν οι ανασχηματισμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και απέτυχε στον ανασχηματισμό εδώ. Και η κυρία Μέρκελ βεβαίω ε, ε, αποφάσισε διότι ό,τι λένε οι Γερμανοί γίνεται πράξη στην σύγχρονη Ευρώπη. Τι έχουμε λοιπόν, κύριε Γιούγκερ, είστε πολύ συμπαθητικό, ε, έχετε θαυμάσια αίσθηση του χιούμορ, καλύτερα από τους περισσότερους που έχω συναντήσει στις Βρυξέλλες, αναμφίβολα. Είστε τεχνικός της πολιτικής, τις τελευταίες εβδομάδες, πηγαίνοντας διάφορες πολιτικές ομάδες, καταφέρατε να αλλάζετε λίγο το μήνυμά σας. Είπατε ότι δεν πιστεύετε στις ΗΠΑ της Ευρώπης, ότι δεν πιστεύετε σε κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που είπατε. Και σήμερα το αποδείξατε. Αποδείξατε ότι εμένετε στις ιδέες της παλιάς Ευρώπης. Μιλήσατε για τον κύριο Ντελόρ, ότι είναι ήρωά σας. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω με βάση τις απόψεις σας. Αλλά επίσης αναφερθήκατε στον κύριο Μητρόν και τον κύριο Κούλ. Είπατε ότι επίσης είναι ήρωές σας. Ε, ο ένας ήταν ε, συνεργάτης ε, κατά την περίοδο της κατοχής και ο άλλος κατηγορήθηκε ότι χρηματίστηκε υπέρ του κόμματός του. Αυτή είναι τα πρότυπά σας σήμερα κύριε Γιούγκερ. Μιλήσατε για την ανάγκη κοινή ε, πολιτική εξωτερικών και ασφάλεια. Μιλήσατε για μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Είναι σαφές ότι θα συνεχίσετε την πορεία συγκέντρωσης εξουσιών, συγκεντρωτισμού εξουσιών. Και αυτό είναι αυτονόητο, γιατί έχετε παίξει ρόλο κλειδί σε αυτή τη διαδικασία συγκεντρωτισμού που έχει αντιμετωπίσει τη δημοκρατία με ηθελημένη περιφρόνηση. Αναφερθήκατε στο γαλλικό δημοψήφισμα για το Σύνταγμα. Ε. Είπατε, αν είναι ναι θα πούμε βεβαίω συνεχίζουμε και αν είναι όχι θα συνεχίσουμε επίσης. Αυτά είναι σοβαρές δημοκρατικές πεπιθήσει. Και η αφοσίωσή σα βασίζεται στο ότι θεωρείτε ότι δεν μπορεί να αναστραφεί. Και είπατε επίσης ότι όταν γίνονται σοβαρά τα πράγματα πρέπει να ε, πείτε ψέματα. Είστε λοιπόν ε, καλός ψήφισε για πολλού εδώ μέσα και αναμφίβολα θα εκλεγείτε αλλά μα ζητάτε να ψηφίσουμε σε αυτόν που είναι ο καλύτερο εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κατεστημένου, που έχει συμμετάσχει σε όλε τι μηχανογραφίε, όλε τι συνωμοσίε και κλεισμένων των θυρών. Και θέλω να πω ότι ο βάδο μου θα σα καταψηφίσει δεν θέλουμε να συνεχιστεί η κατάσταση όπω είναι, θέλουμε ουσιώδη αλλαγή. Στο τέλο τη ομιλία σα είπατε ότι τώρα δεν θέλουμε να κάνουμε επανάσταση, δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Μα έχει υπάρξει επανάσταση ή καλύτερα πραξικόπημα σε σχέση με την δημοκρατία στα εθνικά κράτη. Χωρίς να το, κανείς δεν το πήρε είδηση. Κανείς δεν το πήρε είδηση. Τι υπέστησαν. Αυτές οι εκλογές σε αυτές τις εκλογές μπορεί να μην πήραμε ακόμη οι ευρωσκεπτικιστές την πλειοψηφία αλλά μην νομίζετε ότι θα τα πάμε καλύτερα γιατί η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών τη Ευρώπη δεν θέλουν ένα ευρωπαϊκό κράτος, δεν θέλουν τη σημαία, δεν θέλουν εσάς ω ηγέτη, δεν θέλουν έναν ευρωπαϊκό εθνικό ύμνο. Βεβαίω θα εκλεγείτε και εγώ θα χαρώ να τσακώνουμε μαζί σα την επόμενη θητεία. Για τους μη εγγεγραμμένους τώρα, το λόγο έχει η κυρία Λεπέν. Η κυρία Λεπέν παρακαλώ έχει ήδη λάβει το λόγο. Παρακαλώ καθίστε. Η κυρία Λεπέν έχει το λόγο. Παρακαλώ συνεχίστε κυρία Λεπέν. Παρακαλώ καθίστε δεν έχετε το λόγο κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, καθίστε, δεν έχετε το λόγο. Τον έχει η κυρία Λουπέν. Παρακαλώ, κυρία Λουπέν. Στις 25 Μαΐου Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ σταματήστε να παρενοχλείτε και τελειώς θα αναγκαστώ να σας εκδιώξω. Ως εκπρόσωπο, Τελευταία φορά σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε, παρακαλώ Παρακαλώ να αποχωρήσει ο συνάδελφος από την αίθουσα. Παρακαλώ να εξέλθετε της αίθουσας. Βοηθήστε τον να εξέλθει. Σας παρακαλώ να εξέλθετε από την αίθουσα. Σας παρακαλώ οδηγήστε τον συνάδελφο εκτός αιθούς. Σας παρακαλώ να εξέλθετε της αιθούσεις. Στις 25 Μισό λεπτό κύριε Λεπέν. Μισό λεπτό κύριε Λεπέν. Μισό κύριε Λεπέν. Κύριε συνάδελφε Παπαδάκη, σας παρακαλώ να εξέλθετε τις αιθούσεις. Δεν μπορείτε να ενοχλείτε την εξαγωγή της Ολομέλειας με αυτόν τον τρόπο. Παρακαλώ να αποχωρήσετε. Μπορείτε να επανέλθετε κατά την ψηφοφορία, αλλά σας αποβάλλω τις αιθούσεις. Yeah. Okay, vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λεπέν, έχει το λόγο. Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ Πρόεδρο. Στις 27 Μαΐου η ψήφος των λαών της Ευρώπης άρχισε να ξυπνά την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Γάλλοι πολίτες αποφάσισαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αγαπητοί συνάδελφοι δεν σας αρέσουν αυτά που λέω Έστειλαν λοιπόν το μήνυμα που λέει όχι στην Ευρώπη των Βρυξελών, όχι στην απαγωγή της δημοκρατίας, όχι στη βλακεία των πολιτικών λιτότητας, όχι στη μαζική οργανωμένη μετανάστευση, όχι στην απίσχναση των εθνικών μας ταυτοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεφύγει, είναι ένα θανατηφόρο πρόγραμμα. Οι λαοί φεύγουν από το στόχο αυτό και οι εκπρόσωποι τους ε, είναι εκπρόσωποι μιας άλλης εποχής. Θέλουν να κρατήσουν μόνο τα πλεονεκτήματά τους. Θέλουν να αυτοσυντηρηθούν αυτοί και το σύστημά τους. Και μας δώσατε σήμερα ένα ακόμη παράδειγμα και υπερασπίζεστε τα συμφέροντα άλλων, όχι των ευρωπαϊκών λαών και αγνοείται ουσιαστικά το δημοκρατικό μήνυμα που έστειλαν οι λαοί της Ευρώπης. Οι σοσιαλιστές και οι υπόλοιποι στην ουσία δεν είναι παρά μόνο μισθοφόροι. Το μόνο που έκαναν αμέσως άρχισαν να μοιράζουν τις θέσεις. Αρνούμενοι φυσικά την λαϊκή ψήφο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τους σοσιαλιστές ανάμεσα στο UNP δηλαδή και το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να μιλήσω με γαλλικού όρους άρχισαν να λένε εγώ θα πάρω αυτό, εσύ θα πάρεις το άλλο εγώ θα ψηφίσω υπέρ εδώ, εσύ θα ψηφίσεις υπέρ εκεί και φυσικά ε, μην πιστεύετε ότι ε, διάλεξαν τον Γιούνκερ και όχι τον Σούλτς ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολίτες. Όχι βέβαια, άγνωστοι είναι αυτοί οι δύο, κανείς δεν τους ξέρει. Τίποτα δεν εκπροσωπούν, τίποτα ε, δεν είναι σε θέση να δώσουν. Κύριε Γιούνκερ, ε, φτάσατε πραγματικά στην ηγεσία μιας οργάνωσης την οποία αρνούνται και της οποίας αρνούνται κάθε δημοκρατική νομιμοποίηση οι Γάλλοι πατριώτες. Δεν είστε τίποτα. Και όταν λέτε ότι θέλετε εσείς να καθορίσετε τη ζωή των πολιτών μας, πώς θα το πετύχετε αυτό. Δεν είναι νόμιμες οι αρμοδιότητες σας και οι εξουσίες σας. Υπακούετε στα χρηματοπιστωτικά λόμπι, τα οποία έχουν καταλάβει την έδρα του οργάνου σας και σας διαφθείρουν καθημερινά όλο και περισσότερο. Είστε το αρχέτυπο της άρνησης της δημοκρατίας. Θυμάμαι μια δήλωση που είχατε κάνει το Δεκέμβριο του 1999 σε ένα περιοδικό γερμανικό. Είπατε ότι εμείς λαμβάνουμε αποφάσεις, τις θέτουμε σε εφαρμογή και περιμένουμε λίγο καιρό για να δούμε τι συμβαίνει. Αν δεν ακουστούν πολλές κραυγές και εξεγέρσεις ε, και δεν καταλάβει η πλειοψηφία τι αποφασίσαμε, τότε συνεχίζουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Τι κινησμός, τι ομολογία. Λοιπόν, Εν πάση περιπτώσει ε, είτε ο Μπαρόζο είτε εσείς ε, τα ίδια. Τα ίδια θα καθοδηγούν το παράλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ίδια θα εξακολουθήσουν να αγνοούν τους λαούς, τις χώρες και τον λαό μου, τον μεγάλο γαλλικό λαό. Του δίνουμε λιγότερη δημοκρατία, μεγαλύτερη φτώχεια, μεγαλύτερη ανισότητα, μεγαλύτερη απώλεια εθνικής ταυτότητας ταυτίζεστε, ταυτίζεστε με τη δυστυχία των λαών της Ευρώπης. Ήσασταν υπεύθυνο ενός φορολογικού παραδείσου. Τώρα γίνεστε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οποία προαγωγεί, εν πάση περιπτώσει. Εμείς θα καταπολεμήσουμε την πολιτική σας και εδώ και στις χώρες μας. Εμείς θα καταπολεμήσουμε ενεργητικά την πολιτική σας γιατί πραγματικά βλέπουμε τι μπορεί να κάνει κάθε μια χώρα ξεχωριστά. Οι Γάλλοι πατριώτες είναι οι περισσότεροι τώρα πια, είναι οι περισσότεροι. Έχουν ενθαρρυνθεί από τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών και μπορούν φυσικά να διώξουν την τεχνοκρατική δομή της Επιτροπής σας στην ιστορία και να την ξεχάσουμε πια να γνωρίζετε ότι εμείς οι πατριώτες ευρωβουλευτές θα παρακολουθήσουμε πολύ προσεκτικά τις πράξεις σας. Θα σας καταγγέλουμε συστηματικά. Ιδιαίτερα στον γαλλικό λαό θα καταγγείλουμε το τι απαράδεκτα πράγματα κάνετε εδώ. Είστε υποέλεγχο πλέον κύριε Γιούγκερ. Ε, το σύστημά σας έχει αρχίσει και χάνετε πια. Δεν δέχεστε το μήνυμα των ε, εκλογών. Αλλά εδώ είμαστε σαν πατριώτες για να σας το θυμίζουμε συνεχώς. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Γιούνκερ Παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι πήραν το λόγο εδώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Να ξέρετε ότι άκουσα πολύ προσεκτικά όσα υπόθηκαν. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής μου ζωής, πάντα άκουγα καλά τι έλεγαν τα κοινοβούλια, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βέβαια. Και πάντα παρακολουθούσα τις συζητήσεις σας όλα αυτά τα χρόνια. Συνεπώς σας ευχαριστώ πολύ όλους. Κατάλαβα ότι αν ε, θεωρούσα ότι είναι δικό μου το πρόγραμμα του κάθε κόμματος, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όλοι θα με είχατε ψηφίσει. Εγώ προσπάθησα έχοντας αναλύσει τα διάφορα θέματα, προσπαθώ όσο γίνεται πιο οικουμενικά να τα συμπεριλάβω όλα. Το κοινοβούλιο σας θα ψηφίσει με μυστική ψηφοφορία από ό,τι κατάλαβα. Το σημειώνω γιατί ο κύριος Φάραντς δεν θα ήθελε προφανώς να καταλάβει ποιοι από την ομάδα του με ψηφίζουν και ποιοι όχι. Οπότε με τη μυστική ψηφοφορία αυτό ξεπερνιέται. Η μυστική ψηφοφορία αποτελεί μια υποχώρηση φαντάζομαι που κάνετε προς τον κύριο Φάρετς. Εγώ δεν τα είχα κάνει. Κυρία Λεπέν, σας ευχαριστώ που δεν θα με ψηφίσετε. Δεν θέλω να έχω την αίσθηση ότι με ψηφίζουν αυτοί που απορρίπτουν αυτά τα οποία πιστεύω. Ευχαριστώ κύριε Λεπέν που δεν θα με ψηφίσετε. Ευχαριστώ. βλέπω ότι κατέληξε ζήτηση λίγο νωρίτερα. Ε, Οπότε όλοι οι συνάδελφοι που είναι στα γραφεία του ή στο Bar Luling θα πρέπει να κληθούν να έρθουν ε, στην αίθουσα για να αρχίσει η ψηφοφορία. Διακόπτουμε λοιπόν για 10 λεπτά και θα ξεκινήσει η ψηφοφορία στις 12.25. Παρακαλώ φροντίστε να έρθουν οι συνάδελφοι. Η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 12.25 όποτε, οπότε και θα έχουμε την ψηφοφορία.